i Να ξεκινήσουμε. Έχουμε τον απαραίτητο ρυθμό. Και τώρα να πούμε ότι θα κινηματογραφηθεί η συνεδρίαση και θα μεταδοθεί και μέσω διαδικτύου και να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής ε, πρωινής συνεδρίασης. Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεισηγητές, ο κύριος Γκουελχέρη και ο κύριος Τσαρκόφσκι. Θα γνωρίζετε ότι το σημείο αυτό το εξετάσαμε εδώ και κάποιο αρκετό διάστημα, από τις 4 Οκτωβρίου, με μια ακρόαση με τη συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμόνων και το συζητήσαμε και στις 18 Δεκεμβρίου του περσινού έτους. Την έκθεση που θα εξετάσουμε σήμερα Την έκθεση αυτή την έχουμε συζητήσει στη διάσκεψη των Προέδρων. Οπότε έχουμε χρόνο ως το Σεπτέμβριο, γιατί παρατάθηκε η προθεσμία ολοκληρωσής της. Πρέπει να εξεταστεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013 η έκθεση αυτή. Για την ώρα έχουμε την γλωσσική εκδοχή μόνο στα αγγλικά. Οι υπόλοιπε μεταφράσεις θα είναι έτοιμες νομίζω στις 24 του Ιουλίου. Θα ζητήσω από τις δύο συνεισηγητές να μας παρουσιάσουν το θέμα. Ποιος θα ήθελε το λόγο πρώτος. Sì, poi eh, Gualtieri. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ωραία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από το περιεχόμενο της ακρόασης που αναφέρατε, όπου είδαμε ότι διαφορετικές θεωρήσεις και ερμηνείες της ε, διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης σε σχέση με την ε, νομισματική και οικονομική ένωση και τα θέματα της διακυβέρνησής της, παρουσιάστηκαν σε αυτή την ακρόαση. Μία από τις απόψεις που, παρουσιάστηκαν, που ακούστηκε από τον κύριο Ντυρίς, η οποία φαίνεται να έχει στήριξη από την πολιτική διανόηση, μας λέει ότι λόγω της ασυμματρικής διοργάνωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, κάποια θεσμικά όργανα και ιδίως το Ευρωκοινοβούλιο, δεν μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα εντός της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφήνει ανοιχτό το περιθώριο για να δημιουργηθεί ένα, νέο σώμα ή μια κυβερνητική, ένας διακυβερνητικός φορέας για τη διακυβέρνηση. Εμείς αυτή την προοπτική πρέπει να την εξετάσουμε, διότι βλέπουμε ότι διαφοροποιημένη ολοκλήρωση από ιστορικής άποψης υπήρξε και θα συνεχίσει να είναι ένα από τα έμφυτα χαρακτηριστικά των νομικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέρος της ιστορικής διαδικασίας της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση μπορεί και οφείλει να εξακολουθήσει να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να έχουμε αυθεντική, πλήρη, ολοκληρωμένη νομισματική και οικονομική ένωση εντός των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματική και δημοκρατική η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η έκθεση ξεκινά με κάποιες αιτιολογικές σκέψεις ε, αποσαφενίζοντας τις βασικές έννοιες και δίνοντας την ιστορική παρουσίαση του θέματος, λέγοντας πώς έχει εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση στην ε, ιστορία του, της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείχνει ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση έχει μια διπλή λειτουργία. Να διασφαλίσει την ε, βασική, το βασικό σεβασμό των αρχών με σεβασμό, με τον καθορισμό της ίσης μεταχείρισης για ίσες περιπτώσεις και της άνισης μεταχείρισης για ανώμιες περιπτώσεις. Και μετά καθορίζει τη διαδικασία ολοκλήρωσης ώστε να οριστούν οι λειτουργίες των ομάδων το μελών. Πάντοτε όμως βάσει της αρχής ότι πρώτα πρέπει να γίνεται σεβαστή η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα ότι γίνεται αντιληπτή ως, μέσος, ως μέσο για να υπάρξει περισσότερη ενότητα. Περισσότερη ενότητα λόγω ακριβώς του βασικού, του ουσιαστικού αυτού σεβασμού της αρχής της ποιότητας όπως ορίζεται από τα κείμενα και ως μεγαλύτερη διευρυμένη ενότητα για να μπορέσει εν τέλει να επιτρέψει τη βαθύτερη ολοκλήρωση όλων των χωρών με τις απαραίτητες διαφοροποίησεις για την καθεμία χωρίς να υπονομεύεται η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομιστική της σταθερότητας. Νομίζουμε ότι οι αρχές αυτές συνεχίζουν να ισχύουν και θα πρέπει να αναλύσουμε το πώς μετά από αυτή την ιστορική παρουσίαση. και βλέποντα τις υπάρχουσες ρήτρε για την γεφυροποιημένη ολοκλήρωση που είναι κάμποσε Ξεκινώντας από τα opt-out, τι εξαιρεσει, τα opt-in, τον περιορισμό εδαφικής ε, εφαρμογή, ειδικέ ρήτρε, παρεκκλήσει, ειδικέ ρήτρε για κάτι μέλη που δεν συμμετέχουν στο ευρώ και ούτω καθεξής. Αφού εξετάζονται λοιπόν στις ιδεολογικές σκέψεις όλα αυτά τα στοιχεία, με την ιστορική παρουσίαση και τις αρχές, περνάμε στους ορισμούς. Πρώτα απ' όλα ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση απαιτεί συγκεκριμένε ορισμένες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ενίσχυση των ιδίων πόρων, δημοκρατική λογοδοσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο και ότι αυτά πρέπει να συμβαδίζουν με ενισχυμένη ανάληψη ευθύνη από το Κοινοβούλιο, καθώ και λογοδοσία σε σχέση με τι εθνικέ αρμοδιότητε. Δεν έχουμε εδώ λοιπόν πόλεμο αρμοδιοτήτων με τα εθνικά κοινοβούλια. Του αντίον. Η βασική λοιπόν αρχή εδώ είναι ότι για να είναι πραγματική η οικονομική και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η νομισματική ένωση αποτελεσματική και δημοκρατική θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απαιτεί μια κάποια χρήση των μέσων που προσφέρει διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Μετά εξετάζουμε τις διάφορες διαδικασίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υλοποιήσει μια τέτοια διαδικασία. Τίνουμε να προτιμούμε τις γενικές νομοθετικές πράξεις με παρεκκλήσεις και ρήτρες διασφάλισης ε, αντί του 136 της ενισχυμένης συνεργασίας κάτι που θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν οι προηγούμενες επιλογές δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Από την άλλη, δεν θέλουμε υπερβολική προσφυγή σε διεθνείς συμφωνίες για να αποφύγουμε τέτοια αποτελέσματα. Από την άποψη την θεσμική, τονίζουμε κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, Δηλαδή, η υπάρχουσα έλλειψη συμμετρία στο 136 λόγου χάρη και στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου, της ψηφοφορία του Συμβουλίου με διάφορε μεθόδους και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. οι οποίοι βάσει των δικαιωμάτων τους ορίζουν ε, τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να θεωρηθεί ω υπονόμευση της νομιμότητας μιας πράξης που υιοθετείται βάσει αυτών των διαδικασιών, αλλά αντιθέτω, ότι αυτή η έλλειψη συμμετρίας ενισχύει την νομιμότητα. Διότι η ισορροπία μεταξύ της συμμετοχή μόνο των ε, συμμετεχών των κρατών μελών και από την άλλη την εκπροσώπηση όλων των πολιτών, όλων των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό τελικά καταλήγει να δημιουργεί ισορροπία μεταξύ των γενικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ειδικών συμφερόντων όσων συμμετέχουν στους ε, διαφοροποιημένους μηχανισμούς. Η ισορροπία αυτή ενισχύει τελικά την νομιμότητα και δεν την υπονομεύει. Αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι κανείς δεν βρήκε ότι δεν ήταν θεμητός ο κανονισμός του 2 και του 6 που, που εγκρίθηκε βάση, με νομική βάση το 136 και το 121.6%. Ε, Επίσης μεταξετάζουμε τη συνεργασία του Ευρωκοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια, η οποία δεν υποκαθιστά την ανάγκη μεγαλύτερης δημοκρατικής συνομιμότητας και λογοδοσίας για το επίπεδο ανάληψης, λήψης αποφάσεων και το επίπεδο στο οποίο αυτές εφαρμόζονται. Τέλος, το πλέον σημαντικό είναι το πώς μπορούμε να πάμε σε μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση και την ολοκλήρωσή της βάσει των υπαρχουσών συνθήκων και όσων προβλέπουν και στο πρώτο τμήμα της έκθεσης περνάμε στο πολύ ευαίσθητο θέμα της ε, αναθεώρησης των συνθηκών. Εδώ προτείνουμε ενδεχόμενες, πιθανές τέτοιες αλλαγές σε συγκεκριμένα άρθρα λαμβάνοντας ως σημείο αφετηρίας την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και τα ζητήματα που απασχολούν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση με κάποιες θεσμικές αποχρώσεις. Δεν μπορώ να συνοψίσω όλο το περιεχόμενο της πρότασης που γίνεται σε αυτά τα κεφάλαια. Απλώς θα σταθώ στα πλέον σημαντικά και θα ολοκληρώσω. Εξετάζουμε το νέο μοντέλο των μηχανισμών παρέμβασης στο ευρώ, ενός δεσμευτικού μηχανισμού δηλαδή, που είναι ανοιχτό στην εθελούσια συμμετοχή των κρατών μελών. Αυτού του τύπου η ανοιχτή ολοκλήρωση θεωρείται το βέλτιστο πρότυπο, το βέλτιστο μοντέλο, αντί να έχουμε μια ξεχωριστή ανάπτυξη της Ευρωζώνης και της ολοκλήρωσής της. Μετά να πτήσουμε το θέμα του ενίου μηχανισμού ε, διάσωσης ανάλογα με τα όσα ορίζει η, Ευρωπαϊκή, Νομισματική Ένωση βλέπουμε τα προγράμματα των συμβάσεων και το πώς μπορεί να έχουμε ένα πολυεπίπεδο προπολογισμό εντό του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις υπάρχουσες διαδικασίες αναπτύσσουμε την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το Ταμείο Επαναγοράς του Χρέους, με την νομική βάση, τι γίνεται με τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν επινοούμε κάτι καινούριο πάντως. Αντλούμε από τις υπάρχουσες προτάσεις και τα έγγραφα της, τις προτάσεις της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Το τελευταίο τμήμα που αφορά την αλλαγή των συνθήκων υποτίθεται ότι είναι κάτι που θα συζητηθεί στη συνέλευση με συγκεκριμένε τροπολογίες. Απλώς είναι λεπτομερέστερες από ό,τι συνήθως και αναπτύσσουν κάποια στοιχεία που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επόμενη συνέλευση. Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ρόλος του Ταμείου και του Επιτρόπου που είναι επιφορτισμένο με τα θέματα ΕΚΟΦΗΝ, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μείωση της πλειοψηφίας ανάλογα με την ψήφο εμπιστοσύνη και την ψήφο μη εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πώς τι λειτουργίες αναλαμβάνουν για την υλοποίηση οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, το άρθρο 9 και κοινωνικές ρήτρε, οι διαδικασίες για τις οικονομικές πολιτικές και τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες, με το 136, δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες, ένα είδος ρήτρας Μετακίνηση, μετατόπιση από το 136 που επιτρέπει την υιοθέτηση νομικών πράξεων βάσει το 136 και η αλλαγή του 136 σε ένα, ένα είδος ανοιχτού άρθρου όπου μπορεί μια χώρα εκτός ευρώ να προσχωρήσει εφόσον το θέλει. Όλα αυτά λοιπόν είναι τροπολογίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο του 136 και είναι σημαντικές. Επίσης το οικονομικό σκέλος. για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 450 αντί για το κλασικό ή δυνατότητα νομικής βάσης για έναν ε, νοσιακό φόρο ο προπολογισμό βάσει των όσων ορίζουν οι συνθήκε, που εμεί θεωρούμε ότι αυτό ο επίπεδο προπολογισμό μπορεί να καταρτιστεί βάσει τη υπάρχουσα συνθήκη, των υπερξών συνθήκων, και επίση η ε, συζήτηση με το Κοινοβούλιο, εφόσον υπάρξει περίπτωση αλλαγή συνθήκη, και η κύρωση από το 1 πέμπτο των κρατών μελών για κάποιε περιπτώσει, καθώ και η παράταση κάποιων διαδικασιών από τις εξαιρετικές νομοθετικές διαδικασίες σε κλασικές ε, διαδικασίες με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτό είναι περίπου το περιεχόμενο της έκθεσης και θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση με την παρέμβαση του κυρίου Τσαρκόφσκη. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ρομπέρτο παρουσίασε τόσο αναλυτικά την έκθεση Οπότε να πω κάτι για το πλαίσιο και τους στόχους. Όπως όλοι ξέρουμε, η συνθήκη της Λισαβόνας υποτίθεται ότι θα ήταν η τελευταία συνταγματική συνθήκη σε μια αλυσίδα συνθήκων που θα μας έδιναν τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτά είχαμε πει και όταν διαπραγματευόμασταν τη συνθήκη του Άμστερνταμ, τη Νίκαια, αλλά λόγω τη ΩΝΕ και τη οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μεταρρυθμίσει. Και αυτό είναι ο κύριο στόχο μα, γιατί εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη μεταρρυθμίσεων. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην εξετάσουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε γιατί αυτό είναι πάντα το δίδαγμα που βγαίνει ότι μετά την ε, σύναψη μιας συνθήκης εξακολουθούν να παραμένουν αρκετές αδυναμίες και περιθώριο βελτίωσης. Ποιο είναι το γενικότερο λοιπόν πλαίσιο. Όταν προσπαθούσαμε να πουλήσουμε την συνθήκη της Λισαβόνας ε, στην κοινή γνώμη λέγαμε ότι θα ενισχυθεί η κοινοτική μέθοδος αν και κάποια θεσμικά ε, όργανα είχαν αμφιβολίες για την εξέλιξη της ε, κοινοτικής δομής, αλλά λόγω της κρίσης οι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής οικοδόμησης ε, αμφισβητούνται. Κάποιες τάσεις τίνουν προς την διακυβερνητική μέθοδο εκτός των συνθήκων. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, κάποια κράτη-μέλη θέλουν να υπονομεύσουν την κοινωτική μέθοδο. Υπάρχει κίνδυνος κατακαιρματισμού. Αν κάποιοι αποδεχθούν ε, αυτή την θεώρηση που ε, παρουσίασε ο Ρομπέρτο στην αρχή της ομιλίας του. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και νέα θεσμικά όργανα. Δηλαδή να επανέλθουμε στο σχέδιο Φουσέ της δεκαετίας του 60. Εμείς ως ε, ΑΦΚΟ πρέπει να αντιδράσουμε γιατί λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο που δημιουργεί ε, πολλές ανησυχίες. Εντάξει, έχουμε δημιουργήσει συνθήκες και θεσμούς που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε την κρίση και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μην επαναληφθεί. Αλλά ως ΑΦΚΟ πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Υπάρχουν τέσσερις εκθέσεις ε, επιτάπητος η δική μας ασχολείται με τη διαφοροποιημένη ενοποίηση με θεσμικές ε, απόψεις για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση αλλά πηγαίνει και παραπέρα. Θα υπάρξει και μία έκθεση για το Συμβούλιο για την αποτίμηση της συνθήκης της Λισαβόνας και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτές είναι οι τέσσερις εκθέσεις που αντιμετωπίζουν τις μελλοντικές προκλήσεις, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρξει ε, σαφής διαχωρισμός μεταξύ των τεσσάρων εκθέσεων. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι να διαφυλάξουμε την κοινοτική μέθοδο και τις προόδους ε, που έχει επιτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε σχέση με την ΟΝΕ και την διαφοροποιημένη ενοποίηση. Είδαμε και ποια θέματα προσπαθούσε να προωθήσει το Κοινοβούλιο στο άμεσο παρελθόν και ήμασταν ε, ε αλλά ελπίζουμε όχι υπερβολικά φιλόδοξοι. Αλλά θεωρήσαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο βασικά ζητήματα. Συζήτησα με τον Άντριου στο Twitter γιατί έτσι επικοινωνεί κανείς άμα θέλει να είναι μοντέρνος. Αλλά ε, ο Άντριου ε, μιλούσε για το διαχωρισμό μεταξύ εθνικής και ομοσπονδιακής λύσης. Κοιτάξτε, εγώ είμαι τόσο ιδιόρυθμος όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι φεντραλιστής και δεν νομίζω ότι είμαι και ανοιχτά εθνικιστής. Αλλά πρέπει να επιληθούν αυτές οι διαφορές ε, στην αντιμετώπιση μας. Η προσέγγισή μας ήταν να διαφυλάξουμε την κοινοτική μέθοδο, να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου και με μερικές ιδιαίτερα φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις Να υλοποιήσουμε λοιπόν κάποιες από τις ιδέες μας. Διότι, ναι μεν ε, προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την ε, διαφοροποιημένη ενοποίηση, αλλά χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να υπάρξει. Ευχαριστώ τον ε, Ρομπέρτο για τη θαυμάσια συνεργασία μας και προσλέπουμε στα σχόλιά σας για τις προτάσεις μας και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ως τις 10 και τέταρτο το πολύ. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας και θα ακολουθήσω το κριτήριο που εύστοχα το πρότεινε ο Αντιπρόεδρος Κόξ. Χθες θα δώσουμε το λόγο πρώτα λοιπόν στους χειώδεις εισηγητές. Πρώτα απ' όλα η Αντιπρόεδρος Γκουρμάη. Thank you very much, dear Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να καλωσορίσω καταρχήν τους δύο συναδέλφους από Κροατία. Ήμουν ε, παρούσα στο άνοιγμα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κροατία. Ελπίζω ότι θα βράσετε τη συμμετοχή σας εδώ και βεβαίως ε, χαίρομαι όταν έχουμε νέα μέλη στην Επιτροπή μας. Ας ε, έρθουμε όμω τώρα στη δουλειά των δύο συναδέλφων. Καταρχήν η συνεργασία ήταν επαγγελματική πραγματικά μεταξύ εισηγητή και συνεισηγητή των δύο συνεισηγητών και δείχνει αυτό την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, αφορά τα βασικά ζητήματα διακυβέρνηση όπως τα ονομάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δι τις προκλήσεις που έχουν σχέση με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την συναρμογή μεταξύ αυτών των, των μελών και των υπολείπων και αφορά και τους άλλους μηχανισμούς εργασίας. Οι δύο συνεισηγητές ε, προέρχονται από τα νέα και τα παλιά κρατημέλη, αυτά που ανήκουν στην ε, ΟΝΕ και αυτά που δεν ανήκουν. Και αυτό είναι σημαντικό. Και θίγουν, όπως είπα, σημαντικά τα σημαντικότερα ζητήματα προκειμένου. Η διαφοροποίηση στη διαδίκηση ολοκλήρωση είναι αναπόφευκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και αυτό είναι και κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα κράτη-μέλη της ε, ΟΝΕ. Από την άλλη μεριά, η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, πρέπει να σε σε αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά χωρί δημοκρατικέ διασφαλίσει. και θέλω να επιμείνω από αυτού. Χρειάζεται διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία και πολιτικός έλεγχος. Συμφωνώ απολύτω με το σχολείο τη έκθεση, όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν θα λειτουργεί ικανοποιητικά η Ένωση αν οι πολίτε δεν γνωρίζουν ποιο είναι υπόλογο. για τη μία την άλλη απόφαση και όταν δεν υπάρχει επαρκής δημοκρατικός έλεγχος. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα σε αυτούς τους τομείς. Συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών οφείλει βεβαίως να διδραματίσει πλήρως τον όρο. του. Την άλλη μεριά πρέπει να συνεργαστεί περαιτέρω με τα εθνικά κοινοβούλια. Παρά τις προσπάθειες στα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος μας ε, μόλις ε, επέστρεψε από την Λιθουανία που είχε μια σύσκεψη αυτή το βράδυ. Η συνεργασία αυτή λοιπόν έλεγα ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Όσον αφορά τις διάφορες προτάσεις τώρα για τις τροποποίησεις της συνθήκης με τις οποίες μιλάτε στην εκθέση πιστεύω ότι η εκθέση περιέχει σημαντικές ιδέες, όπως για παράδειγμα την κοινωνική ρήτρα ή τη ρητρεπιτήρηση του προπολισμού. Η κρίση βεβαίω και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση τη, καθώ και οι σχετικέ ε, συζητήσει τα τελευταία χρόνια συντείνουν προ την ενίσχυση ακριβώ τη εσωτερική λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την εξαιρετική συνεργασία. Πώς Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο συνεισηγητές. Το αποτέλεσμα της εργασίας των οποίων είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στην συζήτηση αυτή στο Κοινοβούλιο αλλά και αλλού. Καθώς προχωρούμε προς τα εμπρός και εν ώψη μιας νέας σύμβασης. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να αμφισβητήσουμε την καθιστική ε, τάξη και να ενισχύσουμε την κοινοτική μέθοδο και να επεκτείνουμε την εφαρμογή της. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι εξαιρετική, εστιάζεται στα θέματα που αφορούν την ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς βρισκόμαστε στην ε, διαδικασία ε, δημοσιονομικής εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει όμως να αγρώμε παράλληλα και τις εξελίξεις με τη μορφή διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης σε άλλους τομείς. Στο προημείο Βλέπω ότι γίνεται αναφορά και στα θέματα δικαιοσύνη και εξωτερικών υποθέσεων. Και εκεί γίνεται αναφορά σε μεταβλητή γεωμετρία, επίση τα θέματα ΚΕΠΑ και ΚΕΠΑ. και όσον αφορά τη δυνατότητα σε εργατικών σχηματισμών κρατών μελών να αναλαμβάνουν ειδικού ρόλους και αποστολές. Ή, επίσης, να δημιουργούν ε, μόνιμους μηχανισμούς συνεργασίας. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συνολικής εικόνας. Θα ήθελα να καταγράψουμε κάποιο τρόπο το τι έφερε η Λισαβόνα στην διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ε, αυτοεξαιρέσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Εν πάση περιπτώσει, το κύριο πιάτο για σήμερα βεβαίω είναι η Ιωνέ και χαίρομαι διότι προειδοποιείται εδώ για τους κινδύνους της διακυβερνητικής πλέον εξεργασίας μέσω της ε, επέκτασης της συνθήκης ε, για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα καταλήξει σε μια σύμβαση μεταξύ κρατών μελών και θα αποτελέσει και τον βασικό τρόπο διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Εάν ε, όντως προχωρήσουμε έτσι, νομίζω θα αποτύχουμε και έχει μεγάλη σημασία το Κοινοβούλιο να καταθέσει τη θέση του περίφραστα για το θέμα αυτό. Πιστεύω επίσης ότι οι θέσει σχετικά με τον συνδυασμό της ενισχυμένης συνεργασίας και της ε, αξιοποίησης του 352 και του, και του άρθρου 136 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Επίσης έχετε δίκιο. Όσο αφορά την άλλη θέση σας, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να οργανωθεί καλύτερα για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα, πιο αποτελεσματικά ακριβώς αυτή η πολυεπίπεδη εσωτερική οργάνωση και διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πιστεύω ότι στην ε, πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία θα ήταν λάθος να ευνοήσουμε την αποσπασματική προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Με πέρα της ε, μάθησης όσον αφορά την ε, Δημοσιονομική Ένωση, αλλά το πώ θα γίνει αυτό στο Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ένα εσωτερικό θέμα του Κοινοβουλίου. Επίση, δεν ξέρω αν έχουμε λόγο εξ αρχή να δώσουμε όλου του ορισμού. γιατί υπάρχει μια σάφεια προς τους όρους ε, Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, επίπεδοι Ευρώπη, οι μαλτιτήρε στα αγγλικά πολλών διαζωμάτων. Και πρέπει να εξηγήσουμε κάποια στιγμή τι σημαίνει ο κάθε όρος. Τι σημαίνουν αυτέ τι τρει ε, έννοιε. Και οι τρεις όροι μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας της ολοκλήρωσης και οι τρεις προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ε, βελτίωση της διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά συνδέονται μεταξύ τους, όμως πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να ξεχωρίσουμε και να ορίσουμε αυτές τις τρεις έννοιες. Επίσης, στην παράγραφο 50, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, αναφέρεστε στην πολιτική γειτονία. Όμως εξελίσσεται και μια παράλληλη συζήτηση αυτή τη στιγμή και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να πω, σχετικά με την αναθεώρηση των όρων συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να αριθμιστεί επισήμω επισήμως με μια μορφή σύνδεση σε κάποιε τομεί. Α το δούμε γι' αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να λύσουμε περισσότερο τα ζητήματα που θίγει η έκθεση. Τέλος. Και προς το παρόν, γιατί είναι πολλά τα θέματα βεβαίως που θίγει η έκθεση, χρειάζεται περαιτέρω σκέψη για όλα αυτά. Στη φάση αυτή λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αναλογιστούμε και την επίπτωση αυτής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στο Δικαστήριο. Γι' αυτό δεν λέτε στην έκθεσή σας. Αν θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε περαιτέρω τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, τη διαφοροποιημένη πορεία προς την ολοκλήρωση, τότε πρέπει να αναλογιστούμε και τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά και στα τρία όργανα που προανέφερα στα τρία άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα οφείλουμε να αναφερθούμε στο ζήτημα. Ίσως δεν είναι η έκθεση αυτή ο κατάλληλο χώρος. Ίσως είναι και πολύ νωρί να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Σύμφωνα με τον Ραφαέλ ότι υπάρχουν και άλλες εκθέσεις που εξελίσσονται στη στιγμή, Λαμασούρ, Ραντζέλ και κάποιους άλλους συνάδελφους των οποίων ξεχνώ αυτή τη στιγμή. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς τους δύο εισηγητές για αυτήν την ε, αναλυτική ε, πρόταση που κάνουν, που περιέχει πολλές προτάσεις. Είναι μια πολύ καλή βάση για αυτή τη σημαντική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε λόγω του αυξανόμενου κατακαιρματισμού της Ένωσης, λόγω του ότι η Ένωση ξεχνάει παραμελεί ή αγνοεί όλο και περισσότερο την κοινοτική μέθοδο και στρέφεται όλο και περισσότερο προς ε, τον ε, διακυβερνητικό δρόμο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να διαφυλάξουμε την κοινωτική μέθοδο και άρα την ίδια την Ένωση και τη Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, μεν, δεν είχα πολύ χρόνο να μελετήσω την ε, έκθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό έγγραφο, αλλά μαζί με τις ευχαριστίες θα ήθελα να κάνω και κάποιες επικρίσεις. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι η πιο σημαντική που διεξάγεται για όλη την ε, νομοθετική περίοδο στην Επιτροπή μας. Περιέχουν, ε, περιέχονται πολλά θέματα για την Ένωση, τις συνθήκες, τις προτάσεις ε, για την ισχύουσα συνθήκη. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση αυτή να γίνει σε βάθος. Να μην αποφασίσουμε στα γρήγορα, χωρίς επαρκή συζήτηση. Χρειάζεται λοιπόν αναλυτική συζήτηση, σε βάθος συζήτηση και αν καταλαβαίνω καλά το άτυπο χρονοδιάγραμμα που συζητήσαμε, δεν θα έχουμε χρόνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Πριν λοιπόν πω δύο λόγια για το περιεχόμενο, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τρόπο ούτω ώστε η Επιτροπή μας να συζητήσει αυτό το θέμα στον αναγκαίο βάθος ε, με την αναγκαία ποιότητα. Δεν έχει καμία έννοια να συζητήσουμε την ε, έκθεση αν δεν την έχουν ε, μελετήσει τα μέλη της Επιτροπής και μετά που θα τη μελετήσουμε μπορεί ξαφνικά να μην έχουμε χρόνο για να τη συζητήσουμε. Δεν μπόρεσα λοιπόν ε, να μελετήσω το έγγραφο αναλυτικά, αλλά από αυτά που είδα με μια πρώτη ματιά που έριξα, βλέπω ότι πρέπει να ενισχυθεί η κοινωτική μέθοδος και πρέπει τα διάφορα θεσμικά όργανα να συνδυάσουν περισσότερο τη δράση τους, να βελτιώσουν τη συνεργασία τους, να δεθούν περισσότερο το ένα με το άλλο. Όμως, με αυτά μεν συμφωνώ, αλλά όμως, ε, όπως ε, και όλα τα μέλη της Επιτροπής, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο με την ησυχία μου και σε βάθος να μελετήσω το θέμα αυτό. Χαιρετίζω τις προτάσεις για την περαιτέρω επέκταση της πολιτικής γειτονίας, να υπάρξει δηλαδή στενότερη συνεργασία για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Χαιρετίζω επίσης, για παράδειγμα, τις προτάσεις που γίνονται να δοθεί περισσότερη επιρροή στο Κοινοβούλιο στην επιλογή και του Προέδρου και των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης δυνατότητας ε, μέσω διαδικασίας ε, μορφής να απολύονται ε, μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου. Και επίσης, ναι αυτό, ότι πρέπει να έχουμε δυνατότητα λοιπόν να εκφράσουμε τη δυσπιστία μας έναντι ενός ή και περισσότερων μελών της Επιτροπής. Αυτά είναι αυτά που ε, θεωρώ σημαντικά. Ακόμη σημαντικότερες θεωρώ ότι είναι οι προτάσεις που ενισχύουν την Οικονομική και Δημοσιονομική Ένωση, άρα ενισχύουν την δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα ήθελα τώρα όμως να ασχοληθώ με ένα θέμα για το οποίο δεν βλέπω να αναφέρονται αρκετά στο κείμενο Υπάρχουν πολλές άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις που είναι αξιόλογες και πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, το πώς θα συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις, πώς θα προετοιμάσουμε μελλοντικέ τροποποιήσεις των συνθήκων μέσω της έκθεσης αυτής, αυτά θα ήθελα να διατυπωθούν ακόμη πιο εκπεφρασμένα. Αυτό ιδιαίτερα για την συμφωνία για μια Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Αλλά παρακολουθώντας και τη συζήτηση στα κράτη-μέλη και εντός των κυβερνήσεων των κρατών μελών, παρακολουθώ λοιπόν ε, τη συζήτηση αυτή που είναι σημαντική. Και είναι σημαντικό εμείς ως Κοινοβούλιο όταν ε, θέτουμε θέμα συντακτικής συνέλευσης να εξηγούμε και τι εννοούμε. Αυτή η συντακτική συνέλευση δεν πρέπει να είναι ένα σώμα που θα συγκληθεί στα γρήγορα και που θα ήθελε στα γρήγορα απλώς να συνυπογράψει μια ήδη ε, διατυπωμένη, ε, εκπονημένη πρόταση, γιατί όπως ξέρετε ότι στις δύο περιπτώσεις που επιχειρήσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα συντακτικής συνέλευση να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα όργανο που με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, της Κομισιόν και των Κυβερνήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών θα είχε τη δυνατότητα να κάνει μια συζήτηση σε βάθος για την περαιτέρω εξέλιξη της Ένωσης και των συνθήκων, κάτι που για μένα σημαίνει ότι δηλαδή διαπιστώσαμε τα αποτελέσματα αυτών των περιπτώσεων, γιατί μέχρι τώρα οι προσπάθειες ε, απέδειξαν ότι δεν αρκούσε ο χρόνος για να συζητηθούν σημαντικά θέματα και ξέρετε ότι αυτό έγινε και πριν τα δημοψηφίσματα στην Ιρλανδία και την Ολλανδία και Αυτές οι συζητήσεις και τα δημοψηφίσματα απέδειξαν ότι τα θέματα τα οποία δεν πρόλαβαν οι συντακτικέ συνελεύσεις να συζητήσουν, αυτά τα ζητήματα προκάλεσαν προβλήματα μετά στα δημοψηφίσματα. Διότι ορισμένα θέματα είχαν περάσει χωρί να υπάρξει ουσιαστική και κατά την παράθεση συζήτηση. Αν θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε πώ θα εφαρμόσουμε το θέμα αυτό τη συντακτική συνέλευση, με τη δυνατότητα και θα έλεγα με την αναγκαιότητα μετά ενό ευρωπαϊκού δημοψηφίσματο για τα αποτελέσματα της συντακτικής συνέλευσης, τότε η διαδικασία της συντακτικής συνέλευσης πρέπει να είναι τέτοια που να δημιουργεί νομιμοποίηση και να ε, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και για τη διαδικασία και για το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει να υπάρχει επαρκής χρόνος, δημοκρατικές διαδικασίες συνολικά στην συντακτική συνέλευση. Θα πρέπει η συνέλευση να ψηφίζει ολόκληρη για τα αποτελέσματα και όχι μόνο το Προεδρείο και άλλα μερικά θέματα που συζητιούνται για το θέμα της συντακτικής συνέλευσης θεωρώ ότι είναι αναγκαία ούτω ώστε η έκθεσή μας να τα αναφέρει σαφώ. Να αρκεστώ σε αυτά και ελπίζω να μην χρειαστεί στην επόμενη συνέδριασή μας το Σεπτέμβριο χωρίς περαιτέρω σε βάθος συζήτηση να χρειαστεί να ψηφίσουμε. Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε βάθος πριν ψηφίσουμε μια τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χέφνερ. Όπως σωστά θυμήσατε, βάσει απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, θα πρέπει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι τρέχουσες προτάσεις. Άρα γίνεται λίγο δύσκολο να υπάρξει παράταση. Και ούτως ή άλλως έχει γίνει ακρόαση, εξέταση της έκθεσης και των γράφων Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αλλά πρέπει να πιεστούμε τώρα για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σόλτ. Παρακαλώ να είστε σύντομο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, μεν δεν έχουμε χρόνο, αλλά είναι από τι πιο σημαντικέ εκθέσει. αυτή και πρέπει να τι αφιερώσουμε την αναγκαία προσοχή. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ για τι πολλέ προτάσει που περιέχονται στην έκθεση και να πω, ανεξάρτητα από το έγγραφο εργασίες... θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν είναι σωστή η απάντηση αυτή στα ερωτήματα. Γιατί το πρόσφατο σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις ε, της NSA θέτει το ερώτημα σε τι δημοκρατική ε, ζωή λειτουργούμε. Ή είμαστε κυρίαρχοι. Υπάρχουν ε, ακόμη πολίτες, υπάρχουν υπεύθυνοι πολίτες που αντιμετωπίζονται ω ενήλικες που συμμετέχουν στην, στην ε, δημόσια ζωή, που μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Και η πολιτική των κρατών μελών και τη Ένωση μπορεί να επηρεάσει όλα τα θέματα αυτά. Ή είμαστε απλώς ε, μία δομή η ειμαστε απλώ είναι πάνω από τους πολίτες και αποφασίζει για τους πολίτες. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η έκθεση αυτή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προσπαθεί να συνδυάσει ε, όλες τις προσπάθειες ε, που γίνονται από διάφορες επιτροπές, την ΕΚΟΝ κτλ. να πλαισιώσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν μπορούμε να ασχολούμεθα μόνο με τη δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να ασχοληθούμε και με την κοινωνική πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ε, ετοιμότητα των πολιτών να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην πολιτική και να μην υπάρξει περαιτέρω αποξένωση από την διαδικασία λήψη αποφάσεων και του πολίτε. Δεύτερον, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε περαιτέρω αυτόν τον διαφοροποιημένο μηχανισμό ενοποίησης ή πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση και να δούμε τι απαντήσει υπάρχουν από την Ένωση και τα κράτη-μέλη. Διότι το Συμβούλιο δεν έχει καμία εντολή στην ουσία για να πάρει τις αποφάσεις που παίρνει. Το αναφέρει ε, το σημείο 8. Πολύ σωστά το, το, ε, η έκθεσή μας. Διαφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ Ένωση και κρατών μελών. Γιατί επιβάλλεται όλο και περισσότερο η μέθοδος Μέρκελ που όλο και περισσότερο προκαλεί διμεροποίηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγνοεί την κοινοτική μέθοδο. είναι ο... Αυτό είναι το συγκεκριμένο ερώτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτή την έκθεση, τότε πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά που συζητιούνται στην ΕΚΟΝ. Βεβαίως και στην ΕΚΟΝ ε, αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα επικριτικά αυτή η πραγματικότητα. Οπότε, επειδή και εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να μελετήσω το κείμενο αυτό σε βάθος, θα έπρεπε λοιπόν να πω ακόμη να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική που παίρνει το Συμβούλιο να συζητηθεί ευρύτερα στην Ευρώπη στα συνδικάτα. Χρειαζόμαστε την ρήτρα κοινωνικής προόδους, προόδου. ούτως ώστε να έρουμε αυτές τις αντιφάσεις. Δεύτερον, χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένη απάντηση στο πώς θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το πρωτογενές και δευτερογενές ε, δίκαιο. Είπε πολλά και ο συνάδελφος Χέφνα για τη συντακτική συνέλευση, συμφωνώ με τη συνολική προσέγγιση του. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το πώς ακριβώς θα έπρεπε να υπάρξει, τι δικαιώματα, τι τρόπο εργασίας θα έπρεπε να έχει μια τέτοια συντακτική συνέλευση. Και τέλος. Και ο συνάδελφος Ντάφ έχει δίκιο που λέει ότι υπάρχουν ε, πολλοί τομείς όπου και σε άλλους τομείς δεν εφαρμόζεται πλέον η, η κοινοτική μέθοδος. Μίλησε για την ε, πολιτική ασφαλείας, μπορούμε να μιλήσουμε για ε, τα θέματα εσωτερικών. Υπάρχουν πολλές πλευρές που πρέπει οπωσδήποτε να τις ε, ξαναδούμε και πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να εργαστούμε για την περαιτέρω βελτίωση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόλτς. Ο κύριος Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Και μάλιστα πολύ χρήσιμη. Διότι θέτει διαφορετικά αλλά αλληλένδετα ζητήματα σε πολλά επίπεδα και διαστάσεις. Μας δίνει λοιπόν μια γενική εικόνα και μια προοπτική όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αν και δεν είχα χρόνο να εμβαθύνω στα ζητήματα και τις πρακτάσεις τους. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Χέφνερ, ο οποίος είπε ότι είναι λίγος ο χρόνος για τη συζήτηση μιας τόσο σημαντικής εκθέσης. Όμως, να υπογραμμίσω δύο-τρεις σκέψεις που ελπίζω να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την οπτική γωνία των συνεισηγητών. Πρώτον, η προσέγγιση αυτή, στο πλήθος της οποίας δεν θέλουμε να επισημοποιήσουμε, αν θέλετε, την ΩΝΕ. Ναι. Και τώρα να συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε κάθε ώρα και στιγμή ότι μεταξύ τους ρυθμίσεις έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα, δεν νομίζω ότι συμβάλλει στην παγίωση, στην ενίσχυση της ΟΝΕ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν συζητούσαμε με την ε, Τραπεζική Ένωση, μία από τις δικές μου επιδιώξεις ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ενισχυθεί με επιπλέον εξουσίες και αρμοδιότητες. Αυτό ήταν τότε το αντικείμενο. Θέλαμε η Έκτη να γίνει μια πραγματική κεντρική τράπεζα. Αλλά έπρεπε να δώσουμε και ένα κίνητρο στα κρατημέλη εκτός Ευρωζώνης να εισέλθουν. Αν δηλαδή συνεχίζουμε να υποτιμούμε την Ευρωζώνη και τους θεσμούς της, έστω ανεπίσημους, δηλαδή που δεν προβλέπεται στην συνθήκη, τότε αποδυναμώνουμε τα κίνητρα το ευρώ να γίνει κοινωνομισμά όλων. Από στρατηγικής λοιπόν πλευράς αυτό αποτελεί σφάλμα. Σίγουρα δεν ενισχύει την ζώνη του ευρώ. Το αντίθετο κάνει. Γνωρίζω ότι κανείς δεν έχει αυτή την πρώτη αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσουμε να κινούμαστε έτσι, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Δεύτερον, και αυτό είναι και η τελευταία μου παρατήρηση, γιατί ότι ή άλλως ε, τα ζητήματα είναι εξαιρετικά πολύ σύνθετα. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι πρέπει να πούμε δύο λόγια για την τάση προς περισσότερες διακυβερνητικές προσεγγίσεις, τις οποίες επικρίνουμε βεβαίω. Ας προσπαθήσουμε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Εθνικών Δικαστήριων προκειμένου. Συμφωνώ με τον κύριο Μόντι, ο οποίο πέρσι τον Αύγουστο επέκρινε τη Γερμανία συγκεκριμένα, διότι μερικές φορέ επικαλούνται τα κοινοβουλιά τους ή τις αποφάσεις των δικαστηρίων τους για να παρεμβαίνουν ή να επηρεάζουν τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι μια κακή συνήθεια. Ένα από τα πλεονεκτήματα της υποσύτηση έκθεσης είναι ότι θέτει τα ευρωπαϊκές ζητήματα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα εθνικά στο εθνικό. Φυσικά εθνικοί θεσμοί όπως τα δικαστήρια και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν και αυτά λόγο την κατάλληλη στιγμή. Τι έγινε όμως το 2011. Θυμηθείτε. έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δευτέρα και Τρίτη, και διέκοψαν την Τρίτη για να συνεδριάσει η Γερμανική Βουλή και ξανά τα ίδια την Πέμπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα με τις σκανδιναβικές χώρες, όπου Έχω μια συγκεκριμένη περιορισμένη εντολή. Δεν λέω ότι πρέπει να κατεργήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια και δικαστήρια, αλλά να κάνουμε τη δουλειά μα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπω πρέπει και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Και για να πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, θυμηθείτε τι έγινε στην Αγγλική, στην Γαλλική Επανάσταση. Όταν έχουμε ζητήματα τα οποία διαπραγματευόμαστε σε επίπεδο κυβερνήσεων να εμπλέκονται κυβερνήσει. Ναι, έχουν την εντολή του στα κοινοβούλια, έχουν και τον τελικό λόγο. Όμω, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, αν συνεχίσουμε δηλαδή έτσι, θα είναι πρόβλημα. Δηλαδή, τι έγινε με την Αγγλία, τι έγινε με την Ελληνική Επανάσταση. Το θέμα είναι οι εκτελεστικέ εξουσίε να ασκούνται από τα εκτελεστικά όργανα της κυβερνήσης και από τα κοινοβούλια. Λέω λοιπόν ότι χρειάζεται και μια άλλη προσέγγιση την οποία δεν μιλάτε στην εκθεσή σα, Πρέπει να καθίσουμε να δούμε ποιο είναι ο ρόλος και ο, και ο σωστός χρόνος εμπλοκής. Και το πλαίσιο παρέμβαση των εθνικών θεσμών όπω τα δικαστήρια και τα κοινοβούλια και πώς τελικώς συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ανεξαρτήτως του ορισμού του, τι σημαίνει πολυεπίπεδος και, και Αυτά τα δύο θέλω να πω. Το πρώτο λοιπόν επαναλαμβάνω είναι και εν παρενθέσει από πω ότι ιδεολογικά δεν είμαι υπέρ τη προσέγγιση αυτή που υποδημάται η δυσυστασία της, της ζώνης του ευρώ και το δεύτερο είναι να αποφασίσουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή το, και το κατάλληλο πλαίσιο και ο κατάλληλος χρόνος για την εμπλοκή των εθνικών θεσμών στα ευρωπαϊκά. Διότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει μια παραδείγμα εμπλοκική παρεμβολή των εθνικών θεσμών. Φυσικά έχουν το δικαίωμα τη κυρία κάποια στιγμή αργότερα, αφού πάρουμε μια απόφαση. Αλλά όχι κατά τη διάρκεια της λήψη αποφάσεων, γιατί περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει η δουλειά μας είναι δύσκολη από εδώ. Από εδώ και πέρα η έκθεση είναι εξαιρετική και είναι και μια ουσιαστική συμβολή στην περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστούμε, κύριο Μπρόντ. Νομίζω η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση είναι ένα ε, εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην διάλυση. Και αυτό ακούγεται αντιφατικό, αλλά θα μπορούσε να μειωθεί αυτή η τάση διάλυση στα δεδομένα του πλέον, του λιγότερο ενθουσιώδους μέλους που είναι συνήθως το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπειτα η ομοφωνία για την αλλαγή των συνθήκων. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε κατακαιρματισμό και αυτό κανέναν δεν θα χαροποιούσε έτσι δεν είναι. Όπω βλέπουμε από το έγγραφο, υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ μορφέ διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, αλλά τρόπον την θα ήθελα να τα απλουστεύσω τα θέματα για να μπορέσω να τα σχολιάσω. Φαίνεται να υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είτε οι συνθήκη που έχουν ε, συμφωνήσει όλοι, αλλά με κάποιες εξαιρέσεις, κάποιο περιθώριο για κάποιες χώρες και έπειτα οι διεθνείς συμφωνίες, οι εκτός συνθήκων. Όπως η συνθήκη του Μάστριχτ που ήταν ε, ένα καλό παράδειγμα. Από τη μια με το κοινωνικό κεφάλαιο και από την ε, άλλη με τα βασικά άλλα θέματα, τα κοινωτικά. Η, ολοκληρωμέ... η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση μπορεί να είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό, με εξαιρέσει. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Με ιδιωτικέ διμερεί δηλαδή συμφωνίε μεταξύ διαφορετικών χωρών. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει τι χώρε στο να είναι λιγότερο συμμετοχικέ, όπως είπε και ο κύριο Νταφ πολύ σωστά. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που γίνεται. Η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση δεν θα επιτρέψει απλώς και μόνο σε κάποιες χώρες να προσχωρήσουν με αργότερους ρυθμούς ή μπορεί και να αντιστρέψει τη διαδικασία. Ο κ. Κάμερον ισχυρίζεται ότι αυτό είναι εφικτό. Εγώ είμαι ιδιαίτερα καχύποπτος ως άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό λέγεται για κατανάλωση από ένα αφελές και εύπιστο κοινό στη χώρα μας. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εκτελεστικές αποφάσεις ή τις συμφωνίες μέσω συνθήκων και κατά πόσον αυτά ισχύουν όχι για το κοινοβούλιο, κάτι που δεν συμβαίνει. Ο κύριος Νταβ ξέρει ότι αυτό δεν είναι δυνατό βάσει των συνθηκών. Υπάρχει λοιπόν εδώ αντίφαση. Οι βουλευτές από χώρες που έχουν καλύπτονται από εξαίρεση συνεχίζουν να ψηφίζουν για θέματα τα οποία δεν θα ισχύουν για τις χώρες τους, άρα για τους ίδιους. Θα παραμείνω σε αυτά, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ωραία. Επειδή πρέπει να συνεχίσουμε και να ψηφίσουμε, θα έρθει και ο πρόεδρος Μπροκ για την ψηφορία της εκθεσής του, θα έλεγα στους εισηγητές, πριν θα ε, σχολιάσετε και συνοψίσετε για αυτές τις παρατηρήσεις, να δούμε τα διαδικαστικά. Γιατί είδαμε ότι υπάρχει θέμα χρόνου, αλλά έχουμε και τον χρονικό περιορισμό για το τέλος Σεπτεμβρίου. Κύριε Γκουαλτιέρη, πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν είναι συμπερασματική η παρέμβασή μου, είναι για τη διαδικασία. Ναι, ήθελα να συμφωνήσουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και συζήτηση. Και μετά κάνετε τη σύνοψή σα μετά την ψηφοφορία. Ναι, συμφωνώ με τι ανησυχίε που εξέφρασαν ο κ. Χαφνερ και άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι όντω χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, 29 Αυγούστου, για την ε, υποβολή τροπολογιών. Δεν νομίζω θα τα καταφέρουμε. Πρότασή μου λοιπόν είναι, σε πρώτη φάση, να ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων να τους πούμε ευθέω και με κάθε ειλικρίνεια ότι την έκθεση την έχουμε ετοιμάσει. Θεωρητικά μπορούμε να τηρήσουμε την προθεσμία. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναβάλουμε και πάπυρον. Είναι σημαντική η έκθεση, όλοι το γνωρίζουμε και το θέμα αυτό το έχουν ε, τονίσει πολλοί συνάδελφοι. Σας ζητούμε έναν και μόνο μήνα επιπλέον. Παράταση ενός μήνα, ώστε η επόμενη συνάντηση να καλύψει τη συζήτηση και άλλη μία για την ψηφοφορία. Μας είπανε ότι και η Επιτροπή ΙΜΚΟ νομίζω ζήτησε κάτι παρόμοιο, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, αλλά αυτό μπορεί και να μας διευκολύνει αν ληφθεί υπόψη. Υπάρχει προηγούμενο. Συμφωνώ ιδίω διότι κάποια από τα σχόλια που έγιναν για να καλυφθούν και αν θέλουμε εμεί να αντιδράσουμε ως εισηγητές θα χρειαστούν αρκετή δουλειά. Ας το πούμε στη διάσκεψη των Προέδρων, χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα μήνα, διότι η προθεσμία για την υποβολή του υπολογιών θα πρέπει να είναι τον ε, Σεπτέμβριο. Οπότε να έχουμε και άλλη μια ευκαιρία να το συζητήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Αρχέ Σεπτεμβρίου. Και προκειμένου να ψηφίσουμε για τη διαθεσμική συμφωνία του προπολογισμού, θα γίνει και μια επιπλέον ΑΦΚΟ, συνεδρία τη ΑΦΚΟ στις αρχές Οκτωβρίου. Α γίνει λοιπόν, α οριστεί η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μετά τη δεύτερη συζήτηση στα μέσα Σεπτεμβρίου χοντρικά. Allora... Ωραία. Νομίζω και καταλαβαίνω, μου ζητάτε να ζητήσω παράταση. Δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να το κάνω. Μου ακούγεται λογικό. Και μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξή. Παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών από τις 29 Αυγούστου, που σε όλους δεν φαινόταν παραδεκτό, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου για να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου της τροπολογίας, 17 Σεπτεμβρίου ας πούμε και μετά να ψηφίσουμε ενδεχομένω τον Οκτώβριο στη Σύνοδο. Μπορείτε να το δεχτείτε. Ωραία. Για το σημείο λοιπόν αυτό, με το σημείο αυτό ολοκληρώνουμε. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Τσαρκόφη. 9 Σεπτεμβρίου αν γίνεται, όχι 5. 9 αν μπορείτε. 9, 9. Προφανώς αλλά έτσι και να το δούμε. Ε, Κάποιο πρέπει να έχει και χρόνο για να μελετήσει τι τροπολογίε για να μπορέσει να τι συζητήσει. Τέλο πάντων, αν θέλετε 9, 9, ωραία. Κλείνουμε εδώ με το σημείο αυτό. Είστε μάλλον το διακόπτουμε το σημείο αυτό τη ημερήσια διάταξη. ορίζω τον πρόεδρο Και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 9 Πότε θα απαντήσετε. Ε, αμέσως μετά. Μετά τις ψηφοφορίες. Είχε αναβληθεί η ψηφοφορία. Δεν θα ψηφίσουμε το θέμα της έγκρισης, τη διαδικασία έγκρισης. Όχι, έχουμε τον προγραμματισμό πολιτικής και μακροπρόθεσμες Δημοσιονομικής Δημοσιονομική επιπτώσει της δημιουργίας ικανοτήτων. Μετά το ψηφοφορία θα μπορούσατε να παρέμβετε. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν απευθεία στην ψηφοφορία. Εκτό αν ο πρόεδρο Μπρόκ έχει κάποια δήλωση να κάνει. αν δεν έχετε κάτι να πείτε για το θέμα για το οποίο ψηφίζουμε σήμερα, να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Μια σύντομη παρατήρηση όταν περάσουμε στις ε, προφορικές τροπολογίες ε, που έχουν γίνει θα προτείνω μία-δύο ελαφρές αλλαγές. Όταν φτάσουμε σε αυτά τα σημεία θα τις παρουσιάσω. Νομίζω ότι συνολικά θα τα πάμε καλά. Βεβαίως, ε, εάν θέλετε, ε, επειδή θέλω να αναλάβω πλήρως τις ευθύνε μου, μπορώ να απαντήσω και σε ερωτήσει αν υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με το κατάλογο των ψηφοφοριών. Έχετε ερωτήσεις ε, να θέσετε στον ε, συνάδελφο Μπροκ. Όχι, ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε απευθεία λοιπόν και ο κύριος Μπροκ θα μας βοηθήσει ζητώντα το λόγο όταν χρειαστεί να διορθώσει κάποιε προφορικέ τροπολογίε. Ξεκινούμε λοιπόν με τη συμβαστική Α Παράγραφος 2. Υπέρ. Να υψώνετε τα χέρια παρακαλώ. Και κοντράρι. Κατά. 2. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν είναι ασύμβατη, άρα μπορούμε να πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία 2 Τσαρκόφσκι. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δύο ψήφι κατά και δύο αποχές. Καταπίπτει η τροπολογία DAF που συμπεριλαμβανόταν στην συμβαστική και περνάμε στη συμβαστική B. Κύριε Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, ο Σνάλφος Έλλης με ρώτησε αν δεν θα μπορούσαμε να βέρουμε κάποια ευελιξία να βάλουμε να δεσμευθούν με, σε, για κάποια μορφή ε, διοργανική συμφωνία, ούτω ώστε στο τέλο ε, να έχουμε κάποια περισσότερη ευελιξία. Ε, εγώ συμφωνώ. Έχει κανεί αντίρρηση με αυτή την προστίκη; Με συγχωρείτε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ότι δηλαδή θα δεσμευτούμε για κάποιου είδους ο κύριος Μπροκ, ε, δεσμευόμεθα υπέρ κάποιας μορφής διοργανικής συμφωνία. Ο κύριος Νταφ, δεσμευόμαστε για κάποια μορφή. Διοργανικής συμφωνίας. Ναι, λέει ο κύριος Μπροκ. Αυτό πραγματικά δημιουργεί ερωτηματικά, αλλά καλό. Να ψηφίσουμε υπέρ. Υπέρ το χέρι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΣΥ. 4α. Κύριε Μπρόκ, θέλετε πάλι το λόγο. Οι αγγλόφωνοι είπαν να μην βάλουμε ότι πρέπει να ε, διευθύνεται και να επιβλέπεται από την ε, Επιτροπή. Όχι να ε, διευθύνεται και να ελέγχεται, αλλά να κατευθύνεται. Το ΕΣΠΑΣ πρέπει να κατευθύνεται και να ελέγχεται από ένα σώμα με την κατάλληλη σύνθεση κτλ. Εντάξει. Κύριε Ντάφ, συμφωνείτε. Συμφωνούν όλοι λοιπόν και ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, τρεις αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίθηκε η συμβαστική ΣΥ, περνάμε στην τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές όπως και πριν εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές ακριβώς το ίδιο εγκρίνεται καταπίπτει η 7 η οποία δεν ψηφίζεται 8 νταφ υπέρ κατά αποχές δύο αποχές 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ λάθος λάθος λάθος και εκτεμένη ταχύτητα 8, 9, 10 η πρώτη τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δύο μέρες υποθέσεις. Τελική ψηφοφορία τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 19 υπέρ, 2 κατά, 3, εποχές. Το σχέδιο έκθεση συγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μπροκ. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το προηγούμενο σημείο. Και τώρα οι εισηγητές Γκουαλτιέρη και Τσαρκόφσκι μπορούν να συνοψίσουν και να σχολιάσουν τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Ας αντιστρέψουμε τους όλους, ο κύριος Τσαρκός. Mm, well, uh... Πρόεδρε. Δύο λεπτά είναι πολύ. Εν συντομία, σχετικά αφορά τους ορισμούς. Αντρίου, έχει απολύτως δίκιο. Χρειαζόμαστε ορισμούς. Το κάναμε ε, και στο γραφό εργασίας. Κοιτάξτε, η αρχική μας πρόθεση ήταν να αναφέρουμε τη λέξη tier στα αγγλικά παρά level, παρά επίπεδο. Να αναφερθούμε στα επίπεδα λειτουργίας τα θεσμικά και όχι τα εθνικά επίπεδα, δηλαδή επιτροπές, ε, εθνικά κοινοβούλια κλπ. Προτιμάμε το tier στα αγγλικά λοιπόν αντί για τη λέξη level. Και ιδιαίτερα χρειάζεται αυτό ο διαχωρισμό εκεί που συζητούμε τα εσωτερικά των κρατών μελών σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα τη εμπλοκή των εθνικών θεσμών, και εκεί δεν πρέπει να υπάρξει σύγχυση. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπε πάλι ο Αντρίου δεν μπορούμε να διευρύνουμε περαιτέρω την έκθεση, να μιλήσουμε για σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά δικαστήρια. Αλλά αν θέλετε ε, να προσθέσουμε τα θέματα άμυνα, ασφάλεια, ε, δικαιοσύνη, ιστορικών υποθέσεων, να τα αναφέρουμε. Αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το περάσουμε με κάποιε τροπολογίε, να κάποιο να ζητήσει περαιτέρω συζήτηση αυτών των θεμάτων. Τον βάλουμε δύο παραγράφου, δηλαδή αυτό γίνεται στο βαθμό που αποσαφηνίζει Δηλαδή τι άλλο εννοούμε, ποια άλλα παραδείγματα, σε ποιου άλλου τομεί θα μπορούσαμε να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία. Τώρα για τα άλλα, πολλά έχω να πω, δεν έχουμε χρόνο όμω, για τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάποιου τομεί συνεργασία. Σύμφωνοι, Θα τον συζητήσουμε, αλλά θα είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν υπέρ και κατά. Πιστεύω ότι το μήνυμα μας προς το Ηνωμένο Βασιλείο πρέπει να είναι ότι είναι δεν μπορεί να τα όλα δικά σου. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμά μα. Είτε σα ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι όπω είναι και τι θέλετε, ούτω ή άλλως σας επιφυλάξαμε προνομιακή μεταχείριση με τι αυτοεξαίρεσει κλπ. Είτε βγαίνετε εντελώς, αυτοξαιρέστε συνολικά, το οποίο θα έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει. Τώρα οι άλλε συμφωνίες, σχέσεις σύνδεση κλπ. Δεν ξέρω θέλει κάποιο δηλαδή να έχει όλα τα πλεονεκτήματα, αλλά να μην πληρώνει για το κόστο των πολιτικών. Αυτό θα ήταν σαφώ αντιπαραγωγικό όταν έρθει η ώρα του δημοψηφίσματο. Εγώ πιστεύω ότι αν ο βρετανικό λάο αντιμετώπιζε ένα ναι ή ένα όχι, θα έλεγε ναι. Αν του δώσουμε όμω εναλλακτικέ λύσεις, άλλε ενδιάμεσε εναλλακτικέ λύσει, δεν νομίζω ότι δεν προ τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ο πειρασμό, το καταλαβαίνω, να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία μορφών συνεργασία. Αλλά αν υποθέσουμε ότι κάποτε πάμε σε ένα δημοψήφισμα. Πάντω, μια που έχουμε και Βρετανού εδώ, βουλευτέ από όλα τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουμε τι θέλουμε τελικά. Σκαλτιέρη, σύντομα. Ο Ραφαήλ τα είπε όλα. Εγώ απλώ να απαντήσω στον Ραντζέλ για το θέμα τη εντός ευρωπαϊκών υποτίμησης των ρυθμίσεων που χαρακτηρίζουν την Ευρωζώνη. Να το αποσαφηνίσω αυτό. Έχουμε δύο μοντέλα. Δύο μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν στις συνθήκες για τα ζητήματα αυτά. Το ένα μοντέλο είναι το μοντέλο ECOFIN, το οποίο συνεδριάζει με όλα τα μέλη, αλλά το οποίο όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε τα θέματα της Ευρωζώνης, να γίνει η επίκληση του 139. Τότε τα άλλα μέλη δεν ψηφίζουν. Πρόκειται για θεσμικό όργανο, είναι το Συμβούλιο έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απλώ σε κάποια σύνθεση ψηφίζουν μόνο κάποια μέλη. Το άλλο, η Ευρωζώνη, είναι μια άτυπη ρύθμιση. Και εδώ είναι το παράδοξο, διότι αφενός είναι Ευρωζώνη, είναι εξαιρετικά ισχυρή, όμως δεν μπορεί να λάβει νομοθετικά μέτρα, δεν μπορεί να νομοθετήσει. Και εμεί είμαστε προκειμένου υπέρ του πρώτου μοντέλου. Δεν θέλουμε να διαλύσουμε την, το Eurogroup. Το Eurogroup πρέπει να παραμείνει ω έχει. Ένα τύπο όργανο συζήτηση. Όμω δεν θέλουμε να μεταμορφωθεί σε θεσμικό όργανο το Eurogroup. Γιατί αυτό είναι κατά τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Θέλουμε η διαδικασία λήψη αποφάσεων να παραμείνει ω έχει, να λαμβάνονται η αποφάση του ΕΚΟΦΗΝ με διαφοροποιημένη συμμετοχή στην ψηφορία, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Όποτε είναι απαραίτητο. Όπως δηλαδή γίνεται σήμερα. Όταν ψηφίζουμε λοιπόν με το 136, τότε τα μη μέλη της Ευρωζώνης απλώς δεν ψηφίζουν. Παρευρίσκονται όμως. Παρακάθενται. Δεν χρειάζεται να πούμε βγείτε έξω επειδή ψηφίσουμε. Όχι. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο υπερασπιζόμαστε. Δεν διαλύουμε το Eurogroup την αντίστοιχη σύνοδο κορυφής. Απλώς διαφοροποιείται ο τρόπος ψηφοφορίας μέσα σε ένα επίσημο θεσμικό όργανο που προβλέπεται στη συνθήκη. Αυτό υποστηρίζω εγώ. Τώρα κάποιοι άλλοι διαφωνούν, αλλά αυτή είναι η βασική μας θέση. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης. Και προ τον κύριο Όσον αφορά τις ψηφορίες εδώ στο Κοινοβούλιο, θεωρούμε βασική πρόληψη της συνθήκης, αυτή που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία ασκείται εμέσως στο Συμβούλιο και αμέσως στο Κοινοβούλιο, διότι εκπροσωπούμε αμέσως τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι τα κρατημέλη. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο μπορεί να διαφοροποιηθεί αφού εκπροσωπεί τα κατημελιστή την ψηφορία, ενώ στο κοινοβούλιο αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί εμεί εκπροσωπούμε την Ένωση, τους πολίτες της Ένωσης. Και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν σκεφτόμαστε για τα συμφέροντα αυτών που δεν συμμετέχουν στην διαφοροποιημένη ψηφοφορία. Εμεί θέλουμε να είμαστε μια δημοκρατική εγγύηση, να συνδέσουμε λοιπόν τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και τα γενικότερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται, έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Το νομοθετικό πακέτο Sixpack γι' αυτό ακριβώς ψηφίστηκε. Τώρα, αν κάποια νομοθετικά κείμενα αφορούν μόνο κάποια κρατημέλη, αυτό γίνεται και με τις ψήφους κάποιων μελών που μπορεί να μην τους αφορά το συγκεκριμένο νομοθέτημα, όμως έχουν λάβει υπόψη τους το γενικότερο συμφέρον. Έτσι εξορροπούνται τα συμφέροντα των ΜΕΝ από τα γενικότερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπροκ, ε, βλέποντας την έκφρασή του, που στέλνει πάλι το λόγο, έστω και σύντομα. Σύντομα, βεβαίω. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι στηρίζω την προσέγγιση των κυρίων ε, Γουαλτιέρη και Τσαρκόφσκι. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό στα πλαίσια των ε, θεσμών που έχουμε να υπάρχει η δυνατότητα απόφασης, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άτυπες δυνατότητες. Εάν δώσουμε επίσημες αρμοδιότητες στο Eurogroup με πρόεδρο, με τη δική του διοίκηση θα αρχίσει να αναπτύσσεται με τρόπο που δεν μπορούμε ποτέ να σταματήσουμε. Οπότε δημιουργεί πρόβλημα στην ε, δυνατότητα συνολική λειτουργίας. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίζουμε περίπου ισότιμα τις χώρες που είναι στην Ευρωζώνη και τις χώρες που δεν είναι ακόμη αλλά θέλουν να εισέλθουν. Και εάν θέλουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε ε, όλα τα μέλη της Ένωσης, δεν έχει έννοια να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα. Διότι ένα νέο ε, όργανο με τη δική του δομή ξέρουμε όλοι την ε, πείρα που έχουμε από τις δικής που ποτέ δεν μπορεί να τις ελέγξεις. Προσπαθούμε να συσπυρώσουμε, όχι να διαχωρίσουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν που είναι αρμόδιος οικονομικά και νομισματικά θα μπορούσε να είναι και πρόεδρος ε, της ε, Ευρωζώνης. Όμως αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούν αυτή τη στιγμή οι άλλοι διότι ε, απαγορεύεται από τις συνθήκες. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Πρέπει, είχε πει ο τα όργανα της Ένωσης να έχουν ε, πρωτοποριακό χαρακτήρα. Αυτό πρέπει να έχουμε ως γνώμονα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι οδεύουν προς την ε, σωστή οδό και θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλείνουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον ε, Αντιπροέδρο Λεσκεβίτσιος. Τον παρακαλώ να περιμένει λίγο ακόμη γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε ε, σύντομα μία έκθεση του κυρίου Ταρκόφσκι για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, αλλά παρακαλώ να μας το παρουσιάσει σύντομα. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. κρίνουμε διαθεσμικές ε, συμφωνίες σχετικά με το ΠΔΠ, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το κείμενο το οποίο ε, έχουμε εδώ τις διαθεσμικές συμφωνίες είναι προσωρινό. Η διάσκεψη των Προέδρων πιθανότατα θα λάβει απόφαση να προσωπήσει το ΠΔΠ τον Σεπτέμβριο, το οποίο σημαίνει ότι 4 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να συνδυάσουμε εντάχει για να ψηφίσουμε και εμείς και έχουμε δύο δυνατότητες. Να πούμε ναι ή όχι με την θεσμική συμφωνία ή να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες και να αναλύσουμε την ουσία του πράγματος. Θεωρώ ότι δεν έχουμε χρόνο για ουσιαστική συζήτηση πριν από τις διακοπές και μετά θα βρεθούμε σε μια ειδική κατάσταση. Έχουμε πολιτική συμφωνία για τον προκλήσμα και εμείς θα ψηφίσουμε Σεπτέμβριο. Τώρα χάρη στους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στην διαπραγματεύση και τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Έχουμε συμμετάσχει στην συζήτηση ουσιαστικά, οπότε απλώ να μπορούμε να επικυρώσουμε την διαθέσιμη συμφωνία έτσι όπως κατέληξε. Στην μορφή αυτή βέβαια που είναι προσωρινή, όπως είπα όμως. Είναι πολύ παράξενη αυτή η διαδικασία. Έπρεπε αυτή η απόφαση να είχε ληφθεί λίγους μήνες πριν, σύμφωνα με το πάγιο χρονοδιάγραμμα, το οποίο προβλέπει ότι περνάει το θέμα και από την Επιτροπή μας. Εν πάση περιπτώσει, λάβαμε μέρος μέσω του κ. Λεμασούρ στην διαπραγματεύση αυτή. Είχαμε παρουσία, οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε τελικά. Επισημένοντας λοιπόν το έκτακτο του θέματος, θα πρέπει και εμείς να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Πρέπει να ορίσω μια προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 24 Ιουλίου στη έκτακτη συνεδρίαση της 4 Σεπτεμβρίου να επιτρέψει να περάσουμε στην επίσημη έγκριση. Ευχαριστώ και χαιρετίζω και πάλι τον ε, τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της ε, Λιθουανίας. ο οποίος θα μας παρουσιάσει βάσει της μέσης διαταξής της ε, συνεδρίασής μας τις προτεραιότητες της Προεδρίας του Συμβουλίου της Λιθουανίας. Θα ε, ακούσουμε τον κύριο Λεσκεβίτσιους γιατί ήταν, ε, υπήρχε και η Κόζακ στην, στο Βίλνιους και ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας βρίσκεται εκεί. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα πω δύο λόγια ε, στα λιθουανικά. Ε, είναι ε, μεγάλη τιμή το ότι είμαι εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας που με καλωσορίζετε στην Επιτροπή σας και καλωσορίζω και ένα από τα άτομα ε, για τα, οποία ε, είναι ο λόγος που είμαι εδώ ο πρώην ε, προϊστάμενός μου και καθηγητής μου ο κ. Άλγιντα Τόρνγκας. Θέλω να σας πω μερικά προσωπικά λόγια. μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπική εμπειρία που είχα η οποία είναι ότι η οποία επίσης με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ε, σκεφτείτε ότι το 1987, όταν ήμουν ακόμη φοιτητής, στην Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λιθουανίας, ένας καθηγητής μου με ρώτησε τι θα ήθελες να γίνεις ε, στη ζωή σου, τι θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου. Και εγώ του είπα θέλω να γίνω φιλόσοφος και διπλωμάτης. Εκείνη την εποχή, το 1987, υπήρχε ακόμη η Σοβιετική Ένωση. Και εγώ ήμουν 17 ετών. Ήμουνα στην πρώτη τελευταία τάξη. μια τέτοια απάντηση βέβαια θα μπορούσε να ε, ακουστεί πολύ περίεργη αλλά ε, να που σήμερα είμαι εδώ και τα έχω καταφέρει να είμαι και διπλωμάτης και φιλόσοφος και με τον πρόεδρο Καζίνη συζητήσαμε διάφορα φιλοσοφικά θέματα ήδη και επίσης είμαι και διπλωμάτης όπως είπα οπότε Ε, νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει και τι απόσταση έχει διανύσει έκτοτε η χώρα μου, ούτω ώστε εγώ σήμερα να μπορώ να είμαι παρόν εδώ ε, ενώπιον μιας από τις πιο φιλοσοφικές θα έλεγα επιτροπές του Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Εκτιμώ ιδιαίτερα τις πολύτιμες συναντήσεις ε, στις οποίες συμμετείχα στο Τσασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα και τον Απρίλιο με εσάς κύριε Πρόεδρε με την ε, κυρία Αντιπρόεδρο που δεν είναι παρούσα καθώς και με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων τον κύριο Νταφ τον κύριο Τσασκόφσκι τον κύριο Χάφνερ τον κύριο Γκουαλτιέρη και την κυρία Γιαννάκο. Σήμερα είναι η στιγμή που πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στις συζητήσεις αυτές μια, σε μια πιο αναλυτική συζήτηση με την Επιτροπή σας για θέματα που είναι τεράστια σημασία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν στραφώ στα επιμέρους θέματα, θα ήθελα να θέσω τις προσπάθειές μας ε, και τη συνεργασία μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πρώτον, σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα ε, πιεστικό οικονομικό κλίμα και υπάρχει επίγουσα ανάγκη να ολοκληρώσουμε το νομικό πλαίσιο ...για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε επίσης ε, του χρόνου το Μάιο τις ευρωπαϊκές εκλογές και λίγοι, όχι μόνο οι δικοί σας, αλλά και η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ε, θέτουν τεράστιες πολιτικές και νομοθετικές ευθύνες στους ώμους των ε, αντιστοίχων ε, θεσμικών οργάνων μας. Δεύτερον, έχουν περάσει περίπου τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό ήταν μια ουσιώδη αλλαγή στην νομοθετική διαδικασία τη Ένωση με ιδιαίτερα αυξημένε αρμοδιότητε για το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα συγκεκριμένα. Θέλω ε, να σα ενημερώσω ότι η Λιθουανική Προεδρία καταλαβαίνει και σέβεται τον συνομοθετικό σα ρόλο. Ε, στο τέλο Αυγούστου ο Υπουργό Εξωτερικών ε, θα καλωσορίσει ε, διάφορου από εσά για μια άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στο Βίλνιους. Θα έχουμε εκεί την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερο μαζί σας για το ακόμη δύσκολο σύνολο διοργανικών θεμάτων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε αυτήν την εποχή μετά την ε, αρχή ισχύω τη ε, συνθήκη Λισαβόνα. Και ε, σας σα διαβεβαιώνω ότι αναλαμβάνω αυτό το καθήκον με καλή διάθεση, εμπιστοσύνη και ενεργητικότητα αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσετε κι εσείς πάρα πολύ, γιατί η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή. Είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να είναι ισχυρός εταίρος της Προεδρίας. Η αποτελεσματική, ε, ε, επικοδομητική και συγκεκριμένη συνεργασία μας θα είναι ζωτική σημασία στο επόμενο εξάμεινο. Έχουμε και, οι δύο, και τα δύο όργανα αυτή την ευθύνη έναντι των Ευρωπαίων συμπολιτών μας, ιδιαίτερα φέτος που είναι το έτος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις ε, καταδεικνύουν ότι η Λιθουανοί είναι ε, μεταξύ των πιο ε, ευρέως θετικών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μου έχει επίσης μια πολύ περήφανη προσπάθεια στο παρελθόν ταχεία εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων. Έχουμε το ίδιο πνεύμα που επέτρεψε στη χώρα μας να ανακάμψει τόσο επιτυχώς από την οικονομική κρίση. Έτσι λοιπόν εγώ και οι άλλοι συναδελφοί μου υπουργοί θα αναλάβουμε το καθήκον ηγεσία του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με μια ιδιαίτερη αίσθηση ε, τιμής, υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα αστραφώ σύντομα στη γενική προσέγγιση της Λιθουανικής Προεδρίας. Με βάση τη θαυμάσια εργασία της Ιρλανδικής Προεδρίας και θα ήθελα να αποτίσω φοροτιμή στα ουσιώδη επιτεύγματά της, η Λιθουανική Προεδρία θα ασχοληθεί με τρεις κυρίως άξονες. Θα εργαστούμε για μια αξιόπιστη, αναπτυσσόμενη και Ευρώπη της διαφάνειας. Πρώτα απ' όλα για την αξιοπιστία. Η οικονομική αξιοπιστία ε, συνοδεύεται από την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την δημοσιονομική εξυγένση. Γι' αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εμβάθυνση της ΟΝΕ και την ανάπτυξη ενός ε, συνολικού πλαισίου για μια τραπεζική ένωση. Μια άλλη προτεραιότητα θα είναι νομοθετικές προτάσεις για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση των χρήματο, χρηματαγορών. Ε, ο δεύτερος άξονας μας είναι η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα δημιουργήσει σταθερές θέσεις εργασίας για, για τον ε, πολίτη της Ευρώπης και που θα αυξήσει και την ανταγωνιστικότητά μας. Γι' αυτό θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το Σύμφωνο για Ανάπτυξη και Απασχόληση. Τέλος, είμαστε υπέρ μιας Ευρώπης της διαφάνειας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Ένωση ως συνολικό πρότυπο διαφάνειας και ασφάλειας θεωρούμε ότι η διαφάνεια είναι και στόχος κάθε αλλά και μέσο για την επίτευξη μιας ισχυρότερης και ασφαλέστερης Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο είναι ο παλμός της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεν έχω λοιπόν καμία αμφιβολία όταν υπογραμμίζω την ε, κρίσιμη σημασία της συμμετοχής όλων των ε, πολιτών της Ευρώπης στις κοινοτικές υποθέσεις. Ε, φέτος είναι Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας. Άρα από οποιαδήποτε προτεραιότητα και αν το δούμε, αξιοπιστή, ανάπτυξη, διαφάνεια, πρώτα απ' όλα οι στόχοι αυτοί πρέπει να εξυπηρετούν τους πολίτες μας. Η Λιουθουανική Προεδρία λοιπόν θα επιδιώξει να αυξηθεί η ε, συνειδητοποίηση, ιδιαίτερα μεταξύ των ε, νέων, των κοινών μας αξιών, αλλά και των ε, δικαιωμάτων που απορρέουν από την ενωσιακή ηθαγένεια. Και σίγουρα θα σας χαροποιήσει το ότι με βάση τους στόχους αυτούς η Προεδρία θα αναλάβει μια σειρά εθνικών και διεθνών διοργανώσεων για να ε, γιορτάσουμε το ευρωπαϊκό έτος ε, της Ιθαγένειας μέσω της άμεσης συμμετοχής του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Υπουργείων, των Πανεπιστημίων και άλλων θεσμών. Το Δεκέμβριο θα έχουμε μια διεθνή διάσκεψη για να σημειώσουμε το επίσημο κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Έτους Ιθαγένεια. Τονίζω επίσης ότι ο ρόλο τη Επιτροπής σα είναι ζωτική σημασία στον τομέα των δικαιωμάτων των πολιτών και τη συμμετοχή στην πολιτική δράση. ιδιαίτερη αξία υποδίδω στην πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που ξεκίνησε πέρσι και θέλω να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τις του να ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Διάλογο ενώπιση των ευρωεκλογών του χρόνου. Δύο εκθέσεις πρέπει να αναφερθούν οπωσδήποτε εδώ. Η μία του κυρίου Νταφ για την βελτίωση της οργάνωσης των ε, προσεχών ευρωεκλογών του Μαΐου που ενέκρινε η Ολομέλεια την περσμένη εβδομάδα και άλλη είναι η δική σας κύριε Πρόεδρε που καλεί τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν υποψηφίους για την θέση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δύο αυτές τις εκθέσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της πορείας μας ε, προς τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η Προεδρία επίσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την ε, συμφωνία η οποία επιτευχθεί ταχεία, τόσο όσον αφορά την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως και την ημερομηνία των Ευρωπαϊκών Εκλογών του 2014. Πιστεύω ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζουν την προσήλωση των θεσμικών μας οργάνων να μην φύσουν προσπαθειών ώστε να πετύχουν οι επόμενες εκλογές παρά τις προκλήσεις στο οικονομικό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, δύο λόγια για συγκεκριμένα θέματα επί των οποίων θα εργαστούμε, θα συνεργαστούμε ακόμη καλύτερα κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Πρώτον, πρόταση για το καταστατικό και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι προφανώς βασικοί πρωταγωνιστές της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Αποτελούν ε, ενσάρκωση της δημοκρατικής συμμετοχής και είναι και εργαλείο για να φτάνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο η φωνή και οι ανησυχίε των πολιτών μας. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν τον δημόσιο διάλογο επί ευρωπαϊκών θεμάτων στην Ευρώπη βοηθούν την κοινή γνώμη να προσανατολιστεί. Από τον περσμένο Σεπτέμβριο η Κυπριακή και η Ατλαντική ε, Προεδρία έκαναν πολλές προσπάθειες για να προχωρήσει αυτός ο φάκελος. Η Ιρλανδική Προεδρία δούλεψε πολύ σκληρά για να καταλήξουμε σε ένα λογικό, ισόρροπο και πολιτικά βιώσιμο ψήφισμα για τον χειρισμό του θέματο τη ε, εγγραφή και επαλήθευση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων του, Είναι κρίμα βεβαίω από την άλλη μεριά ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμβαστική λύση. Λόγω του αντιεξόδου η Προεδρία πιστεύει ότι και τα τρία θεσμικά όργανα τώρα πρέπει να σκεφτούν πώ θα βγούμε από το συγκεκριμένο αδιέξοδο. Τέλο, όσον αφορά την ανεξαρτησία τη αρχή εγγραφή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και το πώς θα χειριστούμε το θέμα της α, απόρριψης απογραφής, διαγραφής ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος στην περίπτωση παράβασης ή μη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Στο Στρασβούργο συνθήκαμε με τον Επίτροπο, εσείς κύριε Πρόεδρε, κύριε Κουρμά, κύριε Γεννάκου, για να δούμε τι προοπτικές ανοίγονται όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Όπως γνωρίζετε, η Λιθωνική Προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει τις σχετικές εργασίες με βάση την εντολή του Συμβουλίου, την πρόοδο βεβαίως που σημειώθηκε υπό η Ελληνική Προεδρία και τις ε, εξέλιξης του τριμερούς πολιτικού διαλόγου. Η Προεδρία μας ελπίζει ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο και επί αυτού του θέματος για να εξετάσουμε περαιτέρω και άλλες πτυχές αυτής της πρότασης όπως τα θέματα της χρηματοδότησης το θέμα τη ευρωπαϊκή ταυτότητα αυτών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στο πλαίσιο τη Εθνική νομοθεσία και άλλα συναφή θέματα. Θεωρώ ότι η συνεργασία με το, με Κοινοβούλιο θα είναι εξαιρετική και προσβλέπω και σε καλύτερα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο φάκελο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Ένα άλλο στόχο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κάτι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, εφαρμογή βεβαίως και της εντολής της συνθήκης της Λισαβόνας. Καταλήξαμε και χαίρομαι γι' αυτό σε ένα κείμενο στο Στρασβούργο. Το επόμενο βήμα είναι να δώσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την γνώμη του όσον αφορά τη συμβατότητα του σχεδίου συμφωνία με τι συνθήκε. Πρέπει να συνεχίσουμε με εξίσου ταχύ ρυθμό και προκειμένου η Προεδρία ελπίζει ότι μπορεί να προσβλέπει στην συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να προσχωρήσει το των δυνατών η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνθήκη. Γνωρίζω επίσης την δουλειά Επιτροπής σας όσον αφορά τις εξεταστικές επιτροπές. Ε, αναφέρομαι στην έκθεση Μάρτιν, όπως ονομάζεται. Ξέρω ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και σε τεχνικό επίπεδο και προσβλέπω όπω ε, είπα στο να σημειώσουμε περαιτέρω προδό για το θέμα. Η Προεδρία θα παρακολουθεί στενά κάθε πρόταση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιτυχάνουμε και τους απαραίτητους συμβασμούς ε, επί των εκκρεμών θεμάτων. Ελπίζουμε ιδιαίτερως ότι θα βρεθεί και επί των ε, θεμάτων που είναι τα πιο προβληματικά για τα κρατημέλη και δει όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, τι ακροάσεις ε, συμμετούχων και τις κυρώσεις. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Αυτά είχα να πω σε αυτή τη φάση τουλάχιστον όσον αφορά τις προτεραιότητες της Λιθωνικής Προεδρίας για τους επόμενους έξι μήνες. Είμαι από τους πιο ένθερμους υπερμάχους της επικοδομητικής και στενής εργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσβλέπω, το παραλαμβάνω, σε στενή και συνεργασία κατά τη διάρκεια των έξι προσεχών μηνών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι πλέον στη διαθέσή σας βεβαίως για να ακούσω τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ε, Υπουργέ. Σας αξίζει χειροκρότημα διότι είναι συμβολική σημασία στο γεγονός ότι η Λιθουανία έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λιθουανία είναι μια όχι μεγάλη, μικρή χώρα, αλλά προεδρεύει σε μια στιγμή καθοριστική. Είναι η πρώτη φορά που μια χώρα πρώην Σοβιετική προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αυτό έχει πραγματικά συμβολική αξία. Άξιζε μόνο και μόνο για αυτό το χειροκρότημα. Να δώσω αυτή αμέσω το λόγο στους συναδέλφους και θα έλεγα να ακολουθήσουμε την ε, σειρά της ε, προσχώρηση στα διάφορα κόμματα. Ο κύριος Ταρκόφιας, ξεκινήσει. Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε κάθε τύχη, ιδίως εγώ που προέρχομαι από γείτονα χώρα, και ως νέα κρατημέλη ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να αναλάβει κανείς ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε περίοδο κρίσης. Καλή σας τύχη λοιπόν. Επιπλέον, η Προεδρία σας φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά σε σχέση με προηγούμενες προεδρίες. Εσείς θα ασχοληθείτε με δύο ζητήματα. Την ολοκλήρωση των υποματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον βλέπετε να υπάρχουν δυσκολίες για τη διοργανική συμφωνία, που είναι το δεύτερο θέμα, ή πιστεύετε ότι μετά την πολιτική συμφωνία θα μπορέσουμε να περάσουμε ομαλά στην ε, επόμενη φάση. Και μετά το θέμα είναι τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το θέμα δεν έχει επιληθεί, νομίζαμε ότι επιλύθηκε πλήρω κατά την Ιρλανδική Προεδρία, αλλά δυστυχώ όλοι σφάλαμε. Προσπαθήσαμε όλοι να μετατοπίσουμε κάπω τι θέσει μα προ το κέντρο για να βρεθεί συμβαστική λύση και βρήκαμε καμιά μέση οδό για να συνεννοηθούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο όμω διαφωνεί. Στους τριμερείς διαλόγους είδαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και ήδη έχουμε μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα που αναμένεται δύσκολη. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιες νομίζετε ότι είναι πιθανότητες να υπάρξει ταχεία επίλυση του προβλήματος. Νομίζω, για να συνοψίσω και τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, έχουμε το βασικό πρόβλημα του πώς να προχωρήσουμε διότι αν δούμε τι γίνεται με το status quo και ποιε είναι οι προθέσεις μας, οι επιθυμίες μας, αλλά και αυτές της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, φαίνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι υπεύθυνο για την ε, λήψη των αποφάσεων σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα. Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστέ. και έτσι έχουμε υπόψη το γεγονό ότι το σκηνικό στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το να επιτρέψουμε σε άλλα πολιτικά κόμματα, νέα πολιτικά κόμματα να σχηματιστούν, να, ε, να ε, δεν είναι πολύ απλό και μας κατηγορούν ότι πρέπει να σταματήσουμε να μπλοκάρουμε το σύστημα που συχνά κάνουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να είναι αμερόληπτο και από την, προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου να ενισχύσουμε και την Επιτροπή Σοφών Ανδρών θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τις διάφορες δυσκολίες το ότι τα κάτι μέλη δεν αισθάνονται άνετα όταν μιλάμε για την ε, εγγραφή και την ε, διαπίστευση. Θα πρέπει να επιτρέψουμε η διαδικασία της ε, εγγραφής να είναι σχεδόν αυτόματη και μόνο ορισμένε περιπτώσει να περνούν από τη διαδικασία επαλήθευση. Μάλιστα, θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της Επιτροπής των Σοφών Ανδρών. Αλλά κάποιος θα πρέπει εν τέλει να μπορεί και να είναι επιφορτισμένος με το να λαμβάνει τις πολιτικές αποφάσεις. Άρα πάλι το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι υπεύθυνο, αλλά με τη συμμετοχή του Συμβουλίου. Και όταν ε, μιλάμε για την εγγραφή, θα πρέπει να καταλάβετε και τη δική μας την τοποθέτηση. Ενώ επιτρέπουμε να είναι σχεδόν αυτόματο το σύστημα, θα πρέπει να σκεφτούμε και τη δήλωση του ενός συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος ότι θα συμπεριφερθούν βάσει των αξιών που αναφέρονται στην συνθήκη προκειμένου να κρίνουμε το αν μια τέτοια δήλωση έγινε καλόπιστα, θα πρέπει να μπορούμε να δούμε το καταστατικό του πολιτικού κόμματο στον ιστορικό του κανονισμό και θα ήταν τελείω αντιπαραγωγικό νομίζω για όλου, ιδιαίτερω για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση όπου ένα εγγεγραμμένο κόμμα, ακόμη και με επαρκή τεκμηρίωση, διατυπώνει δηλώσεις που αντίκενται στη συνθήκη. Αυτό θα γελιοποιούσε ολόκληρη τη διαδικασία. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, να πάρει πολιτικές διαστάσεις αυτή η διαδικασία. Είμαστε κατά μια τέτοια τάση, αλλά θα πρέπει να είμαστε και λογικοί. Και όπως είπα, εντάξει, είναι σχεδόν αυτόματη διαδικασία, αλλά τουλάχιστον ας δούμε τα χαρτιά ενός δεδομένου πολιτικού κόμματος και να δούμε κατά πόσο η πολιτική τους δήλωση έχει υπογραφεί καλό, καλή πίστη ή όχι. Ιδάλλως, αυτομάτως θα εγγράφουμε ένα κόμμα που μπορεί στα χαρτιά του να έχει τοποθετηθεί κατά των ε, βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχουμε φανταστεί. Με το που θα ολοκληρώνεται η εγγραφή θα αρχίζουμε την αποεγγραφή. Μην ε, ε, πλήξουμε τη σοβαρότητα και το κύρος ή οδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα. Χρειαζόμαστε λοιπόν από εσά, και αυτό είναι η λέξη κλειδί, χρειαζόμαστε να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει, χρειάζεται κάποιο, για να το πω απλά, στην καθημερινή γλώσσα, θα πρέπει ε, κάποιο να καθίσει τους, τα μέλη του Συμβούλου γύρω από το τραπέζι και να τους αναγκάσει να λάβουν μια απόφαση. Κάποιε φορέ είναι σε δυσχερή θέση και το Κοινοβούλιο και οι διαπραγματευτέ του όταν έχουμε συνομιλίε με το Συμβούλιο, αλλά εδώ έχει υπάρξει προθυμία. Έχει φανεί προθυμία να πάμε προ την κατεύθυνση του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει την εκτίμησή τη γι' αυτό. Προσπαθήσαμε να θέσουμε επιτάπητο μια πραγματική συμβαστική λύση. Αλλά υπάρχουν και κάποιε κόκκινε γραμμέ, υπάρχουν και κάποια απογραφτικό όρια για μα. Εάν θέλετε να κάνετε μια κοροϊδία, μια φάρσα την όλη διαδικασία, δεν έχει πλέον κανένα νόημα και νομίζω ότι το status quo όπως το γνωρίζουμε ούτως ή άλλως πρέπει να αλλάξει. Είμαστε λοιπόν σε μια διάθεση να βρούμε συμβιβασμούς, να βρούμε λύσεις και θα σας εξυπηρετήσουμε, ιδίως σε τεχνικό επίπεδο. Με τις νομικές υπηρεσίες που μπορούν να αρχίσουν να βολιδοσκοπούν και να μελετούν. Όμως από σας Εάν δεν υπάρξει ηγετικό ρόλο, θα είναι δύσκολο να επιλυθεί το πρόβλημα. Διότι σε κάποιε από τι συναντήσει των τριμερών διαλόγων είχαμε την εντύπωση ότι απλώ δεν υπήρχε εντολή. Εντολή από το Συμβούλιο προ την αντιπροσωπεία του για να επιλέξουν τα εκκρεμή ζητήματα. Το πραγματικό λοιπόν πρόβλημα είναι ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ω το δυνατό ταχύτερα. Και αν δούμε το μέλλον και πώ θέλουμε να διοργανώσουμε τι ευρωεκλογέ, που θέλουμε να έχουν περισσότερο ευρωπαϊκή διάσταση, Αυτό είναι ένα θέμα βάσει το οποίο θα κρυθεί η αξιοπιστία μα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώ βλέπετε την κατάσταση στο Συμβούλιο. Έχετε κάποια κοινή θέση, κάποια κοινή γραμμή έστω. Θα μπορούσε και αυτή να συμφιλιώνεται με τι προτάσει που υπάρχουν επιτάπητο. Και τελευταία ερώτηση. Το θέμα τη Ευρωπαϊκή Διάσταση των ευρωεκλογών. Έχουμε μια εξαιρετική έκθεση, την έκθεση του κυρίου Νταφ, η οποία έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, το Σώμα. Και πιστεύουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό το εφαλτήριο του αγώνα που θα δώσουμε για τις ευρωεκλογές. Και αυτό συζητούμε. Βέβαια, εγώ έχω κάπω ε, συνηθίσει σε αυτό, αλλά ποτέ δεν σταματώ να αφνιδιάζομαι. Υπάρχει μια μακρά ιστορία στα του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων που εκπροσωπούμε ότι θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση ευρωεκλογέ και σε αυτές να υπάρξουν και υποψήφοι που θα προταθούν και για τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε οι πολίτες να έχουν και την εντύπωση ότι οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι επίτροποι επηρεάζονται και από αυτούς. Και ότι αυτό έχει και κάποια επίπτωση στο τι αποφάσει λαμβάνονται στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι κάποια κατημερίδια δεν χαίρονται με αυτή την προοπτική και ούτω καθεξή. Αλλά εκεί, σε τι φάση βρισκόμαστε. Μπορείτε να δεχτείτε την πρότασή μας και αν όχι, ποια είναι η συλλογιστική σας. Υπάρχει περιθώριο για συμβασμούς, γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτές οι, εκλογές, αυτές οι μετά τη θέση σε ισχύ της της Λισαβόνας θα πρέπει κάτι διαφορετικό να φέρουν. Ποια είναι λοιπόν η αισθήσή σας για το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Παρόλο που απόφαση ξέρουμε ότι θα ληφθεί στα ύψιστα επίπεδα, πείτε μας ποιες είναι οι γενικές τάσεις στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην επικεφαλής της αντιπροσωπείας, στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σε αυτή την επιτροπή, τον κύριο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω θερμά από πλευράς της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών την Λιθουανική Προεδρία και τον κύριο Λασκεβίτσους και χαιρετίζω και τις ε, παρατηρήσεις του, το πρόγραμμά του. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Τσαρκόφσκι για το θέμα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Τονίζω ότι ναι μεν μπορεί να μην είναι επίσημη αυτή η ε, διαβεβαίωση αλλά ε, είχαμε την εντύπωση ότι είχαμε καταλήξει επί της ουσίας σε πολιτική συμφωνία. Πρέπει να διευκρινιστεί η εντολή του Συμβουλίου και να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε αυτή τη βάση. Ε, υπάρχει αυτή η άτυπη συμφωνία που de facto προέκυψε το τελευταίο τριμερή διάλογο με βάση το ότι η διαδικασία εγγραφής θα ήταν απόλυτα ανεξάρτητη και θα ήταν μια διοικητική διαδικασία, θα γίνεται από το Κοινοβούλιο, αλλά με έναν μη πολιτικό τρόπο θα είναι καθαρά τυπικό το θέμα από μια ειδική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, αλλά η διαδικασία διαγραφής θα γινόταν και με συμμετοχή του Συμβουλίου, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός συναπόφασης, κάποια συνενετική διαδικασία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι η πολιτική βάση της συμφωνίας που τώρα θα πρέπει να επιδιώξουμε να επισημοποιηθεί ε, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση. Είπατε κι εσείς ότι πρέπει οι επόμενες ευρωεκλογέ να γίνουν πιο πολιτικές και το ευρωπαϊκό καθεστώς των πολιτικών κομμάτων είναι σημαντικό στοιχείο γιατί αυτά ακριβώς τα κόμματα θα ορίσουν ε, τους επικεφαλείς ε, των ψηφοδελτίων τους για να παίξουν ε, τον θεσμικό τους ρόλο στη διαδικασία που θα καταλήξει και στην εκλογή του επομένου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, το νομικό λοιπόν, το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς είναι σημαντικό λοιπόν για τον πολιτικό αυτό ρόλο που αναφέρουν και οι συνθήκες. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταβάλλετε όλες τις αναγκαίες προσπάθειες να υπάρξει σαφής εντολή να καταλήξουν διαπραγματεύσεις για τα πολιτικά κόμματα. Επίσης, καλωσορίζω, καλωσορίζω και αυτά που είπατε για τις επόμενες ευρωεκλογές, την έκθεση DAF, την έκθεση Καζίνη, όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε αυτές οι ευρωεκλογές να είναι διαφορετικές. Να αποτελέσουν βήμα προς έναν ουσιοδός ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο και να ενισχύσουν έτσι την δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεση DAF περιέχονται συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που ναι μεν δεν είναι ευθύνη του Συμβουλίου αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να τα στηρίξει πολιτικά η Προεδρία για να αρχίσουμε να συζητάμε το πώς ακριβώς θα τα εφαρμόσουμε. Ε, προσπάθειες ενημέρωσης, δημόσιες συζητήσεις. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε τους πολίτες, να έχει υπόψη του τι επιλογές θα σημαίνει η ψήφος του. Εκεί πρέπει να βοηθήσει και το Συμβούλιο. Θα ήταν ε, ευπρόσδεκτη μια πολιτική ε, όθηση από το Συμβούλιο με βάση και τις συνθήκες. Γιατί ξέρετε, ακούμε από κάποια σημαντικά κράτη-μέλη άλλες φωνές που αμφισβητούν το πώς θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για την επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα οι συνθήκες λένε σαφώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής με βάση την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και η πρόταση αυτή πρέπει να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών και μετά την ε, πρέπουσα διαβούλευση. Και επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τα κράτη-μέλη, φυσικά δεν θα κάνει διαβούλευση με τον εαυτό του, αλλά με τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έρθει να διαβουλευθεί με τα κράτη-μέλη, μα είναι τα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να κάνει διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και με βάση το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης και των εκλογών να προτείνει στο Κοινοβούλιο τον υποψήφιο πρόεδρο της Επιτροπής, τον οποίον θα εκλέξει το Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να επισημοποιηθούν από πολιτική και νομική άποψη και είναι σημαντικό και η Κομισιόν και η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, ε, στηρίξουν όλη αυτή την ε, πραγματικότητα. Δεν θα την έλεγα καν ερμηνεία. Είναι το γράμμα της συνθήκης. Αυτά λοιπόν τα πιο σημαντικά. Αναφέρατε και άλλα. η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε για να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο συναδέλφος Χέφνερ έχει ζητήσει το λόγο, όμως θα ζητήσουμε από τον κύριο Ντάφ να το επιτρέψει, εάν συμφωνεί, διότι πρέπει κάπου να πάει ο κύριος Χέφνερ. Εξ ονόματος, λοιπόν του κυρίου Χέφνερ. Κύριε Ντάφ, μπορείτε να το επιτρέψετε. Ευχαριστούμε. Κύριε Χέφνερ. Uh, ευχαριστώ. Δεν αρμόζει κανείς από εμάς να παίρνει το λόγο πριν από τον κύριο Ντάφ. Αλλά έχει περάσει πολλή ώρα και πρέπει να πάω σε άλλη επιτροπή. Όπου έχω αναλάβει συγκεκριτή σε μια έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Λιγκεβιτσιούς για την εισαγωγική σας ομιλία που ήρθατε εδώ στην αρχή της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ και για, τις προσωπικές, ε, για την προσωπική ποινωνία που είχαμε. Το εκτιμώ. Εύχομαι σε εσά και τη Λιθουανική Προεδρία πραγματικά πολύ καλή τύχη. Για το σημαντικό αλλά και δυσχερές εγχείρημα που έχετε αναλάβει για την Ευρώπη είναι τεράστια πρόκληση σε αυτή την χρονική περίοδο. Διότι είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη, ώστε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κρίση που διαρκεί και σοβεί να περάσει σε μια δημοκρατικότερη, σταθερότερη περίοδο όπου θα μπορέσουμε με τη στήριξη των πολιτών που θα ανακτηθεί, δύο σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και γενικότερα, να προχωρήσουμε. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και πραγματικά σε δύσκολες στιγμές, με πολλές απαιτήσει από όλες τις πλευρές. Μπορούν όμως να γίνουν για να εμπαθύνουμε τη συνεργασία μας, την οικονομική και νομισματική, την φορολογική, την τραπεζική ένωση και όλα αυτά να έρθουν κάτω από την αιγίδα της δημοκρατικής νομιμότητας και ελέγχου, λογοδοσίας. Δηλαδή βάσει της κοινοτικής μεθόδου και όχι εκτός της κοινοτικής μεθόδου. Θα ενισχυθεί η Ευρώπη και η δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε παράλληλα είναι να εντείνουμε τις συζητήσεις στην Ευρώπη, συζητήσεις με τη συμμετοχή των πολιτών ώστε να υπάρξει περισσότερη νομιμοποίηση και καλύτερη προβολή της πολιτικής μας. Η συμμετοχή, το να ακούγεται κανείς, να εκφράζεται, το να συνειδητοποιεί ότι εγώ είμαι μέρος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπει το να αναπτύξει και μια ταυτότητα. Όταν έχει κανείς ε, ένα ρόλο να διδραματίσει δικαίωμα έκφρασης από την Ένωση, τότε καλλιεργείται η ταυτότητα δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να αποδέχεται απλώς αυτά που αποφασίζονται. Οι προτάσεις του μπορεί να επηρεάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εκλογών, μέσω των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών και ίσως και στο μέλλον με νέου είδους ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα μπορεί να αλλάξουν και άλλα τα πράγματα. Ιδίως σε ό,τι αφορά σημαντικές αλλαγές σε συνθήκες. Για τα θέματα τώρα που αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει. Για τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω βρισκόμαστε κοντά στο να εξευρεθεί κάποια λύση. Ένα συμβασμό που θα μπορούσε να βρεθεί και σύντομα μάλιστα. Με αμοιβέ παραχωρήσει από όλε τι πλευρέ. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειε, διότι ο κ. Τσαρκόφσκι είπε πάρα πολλά γι' αυτό. Από να πω ότι δική μας αίσθηση είναι ότι η συμβαστική λύση είναι εφικτό να βρεθεί. Το Κοινοβούλιο αγωνίζεται για να βρεθεί. Το ίδιο και το Συμβούλιο. Ελπίζω. Οπότε νομίζω ότι θα γίνει αυτό και σύντομα. Για την Εξεταστική Επιτροπή, τις Επιτροπές Έρευνας. Πώς να το πω τώρα. Και εδώ μπορεί να βρεθούν ε, συμβαστικές λύσεις, όσο να το αναφέρει αργότερα ο κ. Μάρτιν, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει κάποια μετατόπιση, κάποια μεταβολή στη στάση του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Χρειάζονται αμοιβέ παραχωρήσεις από όλους. Γιατί τέτοιες επιτροπές καλό είναι να συστηθούν και το πλαίσιο ακριβώς αυτού του άμεσα εκλεγμένου δημοκρατικού σώματος, του Ευρωκοινοβουλίου, να μπορούμε να καλέσουμε μάρτυρες, να έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα και πιστήρια, ό,τι χρειάζεται, ώστε μια εξεταστική επιτροπή να αναλάβει πλήρως το ρόλο που της αρμόζει βάσει του χαρακτηρισμού αυτού. Να μην είναι μια ε, κενή προσπάθεια. Η κίνηση λοιπόν αυτή, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, αλλά χρειάζεται η κίνηση να γίνει και εντός του Συμβουλίου. Συζητούμε τώρα το θέμα για τις έδρες των ευρωπαϊκών ε, οργάνων και είναι και αυτό ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Νομίζω λογικό θα ήταν η συζήτηση να ξεκινήσει και στο Συμβούλιο. Ε, ε, με προοπτική το μέλλον ώστε η συζήτηση αυτή να ξεφύγει από εκεί που έχει τώρα παγιδευτεί να είναι συντηγματικού χαρακτήρα η συζήτηση για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου βάσει των όσων έχουν επιτευχθεί με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας όσα ορίζουν ε, τα άρθρα 10 και 11 των συνθήκων πώς θα διαμορφωθούν ε, οι ομαλές σχέσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις συνθήκες εργασίας αυτού του Κοινοβουλίου το τόπο όπου εργαζόμαστε, τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε ακόμα και βρισκόμαστε ακόμα στο έτος των πολιτών. Δεν αξιοποιήσαμε πρακώς αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά έχουμε και μια υποχρέωση να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που βρίσκεται στη διάθεσή μας, για να δουν οι πολίτες ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για αυτούς και χρειαζόμαστε και θέλουμε τη συμμετοχή τους. Ιδίω για τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν έχει ακουστεί αρκετά. Πρέπει να το εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Σας θέλουμε. Θέλουμε τις πρωτοβουλίες σας. Θέλουμε τις προτάσεις σας. Η Ευρώπη είναι ανοιχτή σε αυτά. Να λοιπόν μια ευκαιρία το δεύτερο εξάμενο αυτού του έτους, του έτους των Ευρωπαίων πολιτών και ε, με ε, την προπτική των ευρωεκλογών να δείξει το Συμβούλιο μια στάση ανοίγματο και πλησιάσματος των πολιτών. Όταν μιλάω για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες των πολιτών, πολλά από τα προβλήματα που έχουμε, ακόμη και τα τεχνικά, η διαδικτυακή συλλογή πληροφοριών, έχουν να κάνουν με το τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Όταν αυτός ο κανονισμός ε, προχωρήσει και αρχίσουν και τρομερείς διάλογοι, τι θέλουμε, να έχουμε ένα απλό ευρωπαϊκό έντυπο για να μπορούν να υπογράψουν τις ε, πρωτοβουλίες οι ευρωπαίοι πολίτες μία βασική διεύθυνση με μια απλή υπογραφή. Για κάποιες χώρες όμως απαιτείται και ο τόπος γέννησης και ημερομηνία γέννηση, όπως η Ελλάδα λόγου χάρη. Οι χώρες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν κάποιον χωρίς αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ε, έντυπο. Αυτό δεν πέρασε στο Συμβούλιο. Καταλήξαμε λοιπόν να έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Οπότε αν κανείς προσπαθεί να υπογράψει την πρωτοβουλία, το πρώτο που πρέπει να πει είναι είμαι Λιθουανός ε, πολίτης ή κάτι άλλο, οπότε πηγαίνει στο κατάλληλο έντυπο κάθε φορά, ανάλογα με το ποιανού κράτος είναι πολίτης. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και με το software ε, το, της ε, διαδικτυακής συλλογής και δεν λειτουργεί το software σε όλα τα περιβάλλοντα των όλων των υπολογιστών. Είναι διαφορετικά τα συστήματα μεταξύ των μελών. Το 2012 πριν τεθεί σε ισχύ έπρεπε να δεχτούμε αυτές τις διάφορες απαιτήσει ε, που διαφέρουν μεταξύ τους από κάτω μέλος σε κάτω μέλος. Όταν φτάσουμε όμως στη φάση της αναθεώρησης το 2015 πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο έντυπο, μία ενιαία μορφή, έναν μορφότυπο για τη συλλογή υπογραφών για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Δεν θα καταστεί αυτό εφικτό εάν δεν αρχίσει από τώρα να εργάζεται το Συμβούλιο για να δημιουργήσει τις προποθέσει και να καταλήξουμε σε αυτή την ενιαία μορφή. Σα ζητώ λοιπόν αυτό να το συμπεριλάβετε στην ατζέντα σα στον κατάλογο προτεραιοτήτων και να δώσετε και στους πολίτες αυτό το μήνυμα, ότι μαζί Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θέλουμε να βελτιώσουμε τις πρωτοβουλίε των Ευρωπαίων πολιτών, να γίνουν πιο φιλικέ προς τους Ευρωπαίους πολίτες, πιο πρακτικές και αποτελεσματικές. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Νταφ. Ε, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Εκ μέρους των φιλελευθέρων σας χαιρετίζω. Τα διάφορα εγχειρήματα φεδεραλιστικού χαρακτήρα στην Λιθουανία μας ενδιαφέρουν πολύ εμάς τους ε, φιλελευθέρους. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια εμβάθμισης της ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας συγκυρίας η οποία χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και μεγάλη αστάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα. Σίγουρα έχετε στα χέρια σας ζητήματα τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν ούτε κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας, ούτε της ελληνικής και, με πάση περιπτώσει, όχι πριν τις εκλογές. Πάντως οι δύο προεδρίες, οι δύο επικείμενες προεδρίες θα σημειώσουν πρόοδο επί όλων αυτών των θεμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν η συζήτηση είναι από τους διδόχους ε, μας μετά τις εκλογές. Σύμφωνα απολύτως και υποστηρίζω την έμφαση που δίνεται στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι πολύ πιο σημαντικό το θέμα αυτό από ό,τι οι περισσότεροι εκτιμούν ή φαντάζονται. θα αλλάξει την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεματικά και θα ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του σχετικού χάρτη. Η ομάδα μας και η Επιτροπή μας αποδίδουν ε, μεγάλη σημασία στην εξέλιξη αυτή. Οι συναδελφοί μου μίλησαν βεβαίως για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δεν χρειάζεται να παραλάβω τα σχόλιά τους. Να πω απλώ ότι δεν αξίζει τον κόπο. Θα ήταν μια πολύ κακή ιδέα να καταλήξουμε σε μια κακή συμφωνία όσον αφορά το καταστατικό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Πιστεύω ότι θα άξει τον κόπο να περιμένουμε και το επόμενο κοινοβούλιο για να διατυπωθεί ένα καλύτερο κείμενο σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας όπως το έχει προτείνει και η Κομισιόν. Θα ήθελα πραγματικά να καταλήξουμε έστω και μετά από λίγο χρόνο σε μια πιο ποιοτική συμφωνία σε σχέση με μια κακή συμφωνία από την πίεση του χρόνου. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν στην έκθεση με το όνομά μου η οποία πέρασε από την Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο με σημαντική πλειοψηφία. Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι έχει μεγάλη σημασία τα κράτη-μέλη να διαβάσουν την συνθήκη της Λισαβόνας. Και μία και δύο και περισσότερες φορές. Για να καταλάβουν κάποια στιγμή ότι ο διάδοχος του κυρίου Μπαρόζου πρέπει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκλεγεί. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με υπουργού από διάφορα κρατημέλη, μερικά από αυτά μεγάλα κρατημέλη, και φαίνεται ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς την εξέλιξη αυτή. Από την έκθεση αυτή της περισμένης εβδομάδας να αναφέρω ότι κάποια σημεία αφορούν το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Το θέμα επίσης της συμμετοχής των γυναικών στα ψηφοδέλτια συμμετοχή που πρέπει να ενθαρρύνουμε σε πολλά, όχι στα περισσότερα κράτη-μέλη. Έχουμε μετά το των ονομάτων και των εμβλημάτων των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων όπως θα εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών Τρίτον, έχουμε το αίτημα να δοθούν δυνατότητες δημοσιότητες στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μέσω των ε, κρατικών ραδιοτηλεπτικών σταθμών. Και το θέμα επίσης των προσπαθειών των κρατών μελών να εφαρμόσουν την οδηγία η οποία επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να ψηφίζουν αλλά και να κερδίσουν ψήφοι σε χώρες άλλες από την δική τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορα εμπόδια σε διάφορα κράτη-μέλη ως προς αυτό. Πέραν των συγκεκριμένων εμποδίων υπάρχουν και γραφειοκρατικά εμπόδια και αντίσταση, απροθυμία θα έλεγα από τις διάφορες αρχές, τα κράτη-μέλη. Και όλα αυτά μαζί έχουν ως τελικό αποτέλεσμα να ακυρώνεται το δικαίωμα αυτό των Ευρωπαίων πολιτών να ψηφίζουν και να είναι υποψήφοι στις εκλογές σε χώρες άλλες από αυτές τι στιγμή έχουν τη μόνη διαμονή τους. Πέμπτον, ζητούμε από τα κρατημέλη να διοργανώσουν δημοσίες εκστρατείες για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις εκλογές, για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και τέλος, ζητούμε να μην δημοσιευθεί κανένα επίσημο αποτέλεσμα πριν να κλείσουν οι κάλπες και στο τελευταίο κράτος μέλος που εμπροκειμένο είναι η Πορτογαλία λόγω Αζωρών. που είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πιο κοντά στις Ηνωμένες παρά στην Λιθουανία, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να λεφτεί υπόψη και η διαφορά της ώρας. ώστε να διεξαχθούν ε, οι εκλογές ε, όπως πρέπει. Προσβλέπω επίση την επόμενη Κόζακ στη... στο Όπου ελπίζω θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα ε, πιο άνετα και με τη συμμετοχή των, ευρωπαϊκών, των, των εθνικών κοινοβουλίων. Ευχαριστούμε κύριε Ταφ. Αλλά επειδή δεν θα έχουμε και ε, ατελείωτο χρόνο, διότι στις 12 αρχίζει κοινή συνεδρία, θα πρέπει να αφήσουμε και στον ε, Υπουργό τον ευκαιρία να ε, αποφασίσει. Για την Στοκόλμη θα μιλήσουμε με τις Επιτροπές Λίμπη και Γιούρι. Λοιπόν, εδώ έχουν εγγραφεί κύριο Άγνιου, ε, Άντριου Μπρόγκς και Γκουρμάη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω ισότιμη μεταχείριση. Γιατί πολλοί συνάδελφοι μίλησαν ε, μακρόν. Καλύτερα να λέμε στην αρχή πώ θέλουν να μιλήσουν και να έχει τρία λεπτά ο καθένα. Ε, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Δεν μπορώ να παραχωρήσω σε όλου ε, παραπάνω από τρία λεπτά. Ε, με τη σειρά λοιπόν, δυόμιση. Ο κύριο Άγνιου πρώτο. Uh, Καλημέρα κύριε Ε, εγώ δεν μιλάω ε, επί μακρόν, ε, όπως οι προηγούμενοι, αλλά δεν θα πω πολλά είστε αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τη Λιθουανία. Με βάση τη συνθήκε Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναπτύξει μια κοινή πολιτική ε, εξωτερικών ε, και ασφάλεια. Σαν να ήταν ε, κράτο. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίξουν αυτή την πολιτική με βάση τη συνθήκη. Όταν θα υπάρξει αυτή η κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλεια, δέχεστε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον λιθουανική εξωτερική πολιτική. Και βέβαια ούτε και βρετανική εξωτερική πολιτική και αυτό βεβαίω με ανησυχεί. Άρα, ξέρετε ότι έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών William Hague του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κάποια στιγμή τα επόμενα δύο χρόνια θα τον καλέσει ο Πρωθυπουργό ε, Κάμερον και θα του πει «Κοίταξε, η κυρία Θάτσερ είχε πει Όλοι χρειάζονται έναν ε, Willie. Αλλά εγώ θα χρειαστεί να σε απολύσω. Οι Βρετανικοί συντηρητικοί σήμερα δεν έχουν έρθει. Γιατί μάλλον ε, φοβόνται ε, ότι φοβήθηκαν ότι θα πω κάτι σαν αυτό που είπα τώρα. Εσείς όμως πώς αισθάνεστε. Εσείς οδεύετε προς την απόλυση. Δεν σας ανησυχεί αυτό. Είχα ξεχάσει να πω μεταξύ αυτών που είχαν το λόγο τον κύριο Σόλτ που είχε βγει, για, δύο λεπτά. Σα δίνω όμω τώρα την ευκαιρία. Όπω έδωσε το παράδειγμα ο κύριο Σάκη, να μην με κρηγορήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή του κύριου Υπουργού στα βασικά σημεία της Προεδρίας του. Και εγώ είχα ερωτήσεις για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα συγκεκριμένα. Πώς βλέπετε να συνδέεται το θέμα αυτό με την ε, κάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να το σημείο αναφοράς για την πολιτική πρακτική των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Μιλήσατε για την αξιοπιστία, ότι είναι ουσιώδες ε, στοιχείο που ως ε, Λιθουανική Προεδρία είναι προτεραιότητά σας. για να είμαστε αξιόπιστοι έναντι των πολιτών. Πρέπει να ασχοληθούμε όχι μόνο με τα οικονομικά αλλά και, αλλά και με τα κοινωνικά θέματα σε όλα τα 28 κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η Λιθουανική Προεδρία πώς θα συμβάλλει ούτω ώστε να, να μην εξακολουθήσει να μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών. να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, όταν ε, διαπιστώνουν οι πολίτες ότι λαμβάνονται ενωσιακές αποφάσεις που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των χωρών. Συζητήσαμε σήμερα την έκθεση Γκουαλτιέρη Τσαρκόφσκι. Τι θα κάνει η Λιθουανική Προεδρία ούτως ώστε μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναρχίσει να εκπροσωπεί και να ασχολείται με τα ε, ζωτικά συμφέροντα της Ευρώπης. Έτσι θα πείσουμε τους πολίτες να ασχοληθούν με το πολιτικό γίγνεσθε. Είναι αυτό βασική προϋπόθεση για να επιτύχουν και οι προεκλογές. Πρέπει λοιπόν να δράσει εντόνως η Λιφανική Προεδρία, γιατί αλλιώς ε, θα εξακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αποτυχάνει. Ευχαριστώ κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, απλώς να επικεντρωθώ σε ένα στοιχείο για το ντοσιά μου και για την Εξεταστική Επιτροπή. Θα ξέρετε ότι οι νομικές υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων έχουν εργαστεί σκληρά για να βρουν τεχνική λύση στο θέμα αυτό. Και Έχω σιωπήσει κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας για την ώρα, αλλά πρέπει να προχωρήσει το θέμα, γιατί οι νομικές υπηρεσίες δεν έχουν επιτελέσει ιδιαίτερη πρόοδο. Θέλουμε να περάσει και πάλι στην πολιτική αρένα το θέμα για να γίνει πρόοδος, οπότε ελπίζω η Προεδρία σας να λάβει και να επιληφθεί. Ε, ξέρετε ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια μορφή συμφωνίας, αλλά ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερω για την ουσία του θέματο. Το είπε και ο κ. Χέφνερ και ε, πραγματικά θέλουμε να επιτελεστεί πρόοδο για την πρόσβαση στα ε, έγγραφα για τη διαδικασία τη συναπόφαση. Ιδάλω οτιδήποτε άλλο θα ήταν κενό νοήματο. Θα Ήθελα να θυμίσω στου συναδέλφου σα ότι εδώ και 34 χρόνια από τι πρώτε ευρωεκλογέ μόνο τρει εκδαστικέ επιτροπέ δημιουργήθηκαν για κάποιου ε, ε, συναδέλφου του Συμβούλου που πιστεύουν ότι με την πρώτη ευκαιρία θέλουμε να συστήσουμε μια εκδαστική επιτροπή. Από κοινού λοιπόν συστήνουμε μια επιτροπή, τη συνθέτουμε για να προσπαθήσουμε να βρούμε την αλήθεια σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα με τα απαραίτητα στοιχεία. Τα κράτη-μέλη με τα οποία τα συζήτησα διμερώ αυτό να ξέρουν ότι δεν είμαστε δικαστήριο την αλήθεια προσπαθούμε να διερευνήσουμε. Άλλοι αποφασίζουν μετά τι θα γίνει και τι όχι. Δεν είναι ένδικο μέσο. Δεν έχει σχέση με το κοινοβούλιο αυτό. Θέλουμε να δούμε ζητήματα κακοδιαχείρισης, ε, φωτίζοντας όλες τους τις πλευρές. Όταν έγινε η προηγούμενη έρευνα, είδαμε ότι δεν είχαμε επαρκή στοιχεία για να φτάσουμε στην αλήθεια και τα κάτι μέλη το αναγνώρισαν ε, συμπληρώνοντας το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνοντά του την συνθήκη τη Λισαβόνα. Ξέρουν λοιπόν ότι κάποιε φορέ πρέπει να αναλαμβάνεται δράση για τέτοια θέματα και ξέρω ότι χρειάζεται πολιτική στήριξη εδώ. Η τεχνική δουλειά έχει γίνει. Τώρα έχουμε ενδείξει ότι πολιτική επιθυμία χρειάζεται για να, πολιτική βούληση για να επιτευχθεί η συμφωνία. τίποτα δεν θα γίνει. Το κοινοβούλιο έχει προειδοποιήσει, έχει διαμορφώσει το σύστημα σωστά ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε την αρμοδιότητα να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα, εφόσον δεν υπάρξει δυνατότητα πρόσκλησης μαρτύρων, δεν θα έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ε, κάθε Προεδρία μάλλον χαρακτηρίζεται από τη χώρα την οποία η οποία προεδρεύει. Εδώ όμως εκτός από τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας θέλουμε να έχουμε και συνέχεια πολιτική. Ε, και δεν θέλουμε τα πάντα να καθορίζει η Τρόικα των Προεδριών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδοχή των χωρών, η πιο πρόσφατη, είναι αρκετά αποκαλυπτική. Αυτό το πρόγραμμα, όπω και άλλα, δείχνει τι ίδιε ελλείψει. Ναι, χωρίς να θέλω να είμαι ιδιαίτερα επικριτικός από τη μια ζητά την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ενώ από την άλλη την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα που θα πρέπει να τονωθεί σε περίπτωση κυριαρχών κρατών που είναι μέλη της Ευρωζώνης με κοινό νόμισμα που είναι πολύ ψηλής αξίας για τις οικονομίες τους και έχουν φανεί τώρα, έχει φανεί μέχρι τώρα ότι δεν είναι ανταγωνιστικά. Επίσης για την ανεξαρτησία των αρχών εγγραφής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Μα τι μπορεί να σημαίνει αυτό τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους όπως στο Σύνταγμα του 1936 της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, είναι σαν να γίνεται εγγραφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο, πόσο ελεύθερο μπορεί να είναι τέτοιο πολιτικό σύστημα. Επίσης, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το τι έγινε με τις πρώτες αιτήσει για διαγραφή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συμπιέλευαν στην αίτησή τους τους λόγους για τη διαγραφή. Αυτό δεν είναι σαν να καλούμε τις διοκτικές αρχές και την αστυνομία να δικάσουν ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά να, να ξεχνάμε να πούμε γιατί κατηγορείται η κοινωνία, η ελεύθερη κοινωνία, η ανοιχτή κοινωνία θα πρέπει να επιτρέπει την αντιπαραβολή διαφορετικών απόψεων και την ελευθερία του ε, τη για ομάδες ατόμων. Εάν αυτό δεν επιτρέπεται, μιλάμε για περιορισμό της δημοκρατίας ή και για την απουσία της η εγγραφή των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάτων με διαφορετικού υποψηφίου για την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το ενδιαφέρον. Είναι όμω μια απόπειρα από αυτό το σώμα να, πούν, ε, να πει στου ψηφοφόρου με τι κριτήρια θα πρέπει να ψηφίσουν. Προβλέποντα ιδιαίτερα προνόμια Κάτι που αφορά και την, ε, τις ποσοστώσεις για τις ευρωεκλογέ και το χρόνο κάλυψης στα τηλεοπτικοακουστικά μέσα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με τι κριτήρια θα μπορούν οι πολίτες να λάβουν ελεύθερη απόφαση. Δεν μπορούμε να τους πείσουμε να ψηφίσουν για ένα πολιτικό κόμμα που δεν έχει καθεστώς Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος και του οποίου οι ψηφοφόροι δεν μπορεί να είναι και πρόεδροι, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε ότι και μια τέτοια ψήφος είναι τελείως πεταμένη. Η κυρία Γκουρμάη. Ε, Πρόεδρε. Σίγουρα διαβάσετε το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας, μοιράστηκε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Είναι μια ευκαιρία να το διαβάσουμε όλοι προσεκτικά. Καλό το ίντερνετ, αλλά καλό να διαβάζουμε και μερικά πράγματα στο χαρτί καμιά φορά. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ κύριε Υπουργέ και συγγνώμη για την καθυστερημένη μου άφηξη. Να πω κι εγώ δύο λόγια για την διαπραγμάτευση όσον αφορά το καθεστώ, καταστατικό και την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους. Χαίρομαι που θέλετε πολιτικός και νομικός να προχωρήσετε στο θέμα. Πάντως, να ξέρετε ότι τα μεγάλη πίεση, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν αποτέλεσμα. κάτι που δεν έγινε υπό Ιρλανδική Προεδρία. Το Κοινοβούλιο πάντω και η Επιτροπή έχουν συνεργαστεί πολύ ικανοποιητικά μεταξύ του και με το Συμβούλιο και πιστεύαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά. Και ξαφνικά, ε, δυστυχώ. Διαπιστώσαμε ότι ήταν αδύνατον να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όσον αφορά τη θεσμική πτυχή, εγγραφή, διαγραφή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων κλπ. Οπότε περιμένουμε η Λιθουανική Προεδρία να, κάτι, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο, γιατί σοβεί η δημοκρατική κρίση, η κρίση δημοκρατικών θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δύσκολο να καταλάβει ο κόσμο ε, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε αυτό το οποίο όλοι θέλουμε και αυτοί περιμένουν. Όπως αναφέρατε και εσείς, εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα όπως η διατάξη περί χρηματοδότησης και η σχέση με τις εθνικές ένωμες τάξεις. Οι εντολή που έχουν ε, διάφορες ε, χώρες εξαρτάται και από τις εθνικές ένωμες τάξεις. Σκοντάτε λοιπόν το θέμα στο Συμβούλιο για να κλείσει αυτό το σημαντικό θέμα το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων για να προετοιμαστούμε και καλύτερα εν ώψη της επόμενης φάσης της διαπραγματεύση, όπω ο Ραφάλ και ο Ρομπέρτο, οι εκλεκτοί συναδελφοί, είπαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει προβεί σε παραχωρήσεις σε υποχωρήσεις και έχει στείλει το μήνυμα. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε καμία περίπτωση. Και το αποδείξαμε νομίζω και κατά τη διάρκεια τη διαπραγματεύση πώ βλέπουμε πλέον τη δική σα συμβολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπούζη τη τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σε μας. Ευχαριστώ που καλωσορίζετε τους συναδέλφους και τη χώρα μας. Χαιρετίζω και ευχαριστώ την Λιτσουανική Προεδρία διότι η Λιθουανία είχε την ευκαιρία να μας καλωσορίσει ως το 28ο μέλος της Ένωσης. Την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την Προεδρία, το πρώτο λεπτό, τα μεσάνυχτα της 30 ε, Ιουνίου προς την 1η Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, τι εκπροσωπεί η Ένωση. Μια χώρα που προηγουμένως ανήκε στη Σοβιετική Ένωση χαιρετίζει μια άλλη ε, πρώην κομμουνιστική χώρα και εγώ προσωπικά θέλω να τονίσω ότι το όνειρό σας κύριε Υπουργέ το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα συναντιόμαστε εκεί ακριβώς που θα θέλαμε. Στην πραγμάτωση των ονείρων και των δυο μας. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό σας στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, την, ε, την πρόεδρο σας και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία παρουσίασε θα επιτευχθούν. Ναι, πράγματι. Η σύμπτωση αυτή, η Λιθουανία πρώτη φορά να αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, μια πρώην κομμουνιστική χώρα, mm. με την ταυτόχρονη προσχώρηση της Κροατίας, αυτό τελικά μας φέρνει στην καρδιά ενός θέματος που απασχόλησε την Ιρλανδική Προεδρία. Πολιτική γειτονίας. Ποια θα ήταν δηλαδή η σωστή ισορροπία με άλλες δυνάμεις ε, εξανατολών όπως η Κρουάνια, η Ρωσία. Αλλά τώρα θα δώσουμε χρόνο στον κύριο Λευκοβίτσιο μετά από τις τόσες πολλές παρεμβάσεις που έγιναν για να μας πει τα δικά του σχόλια. Και θα μπορέσουμε την κοινή μας αυτή προσέγγιση να την αναπτύξουμε περαιτέρω και στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. τις προτάσεις επίσης, την καλή σας ε, θέληση και διάθεση να συνεργαστείτε με το Συμβούλιο και με μένα προσωπικά. Να συνεργαστείτε επικοδομητικά. Πριν απαντήσω στις ερωτήσεις σας, και το πόσο πολλοί άριθμες ήσαν δείχνει τη σημασία της Επιτροπής σας και των θεμάτων που μας απασχολούν να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις. Σας ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσω. Θα πρέπει να απαντήσω σε ομάδες ερωτήσεων. Δεν νομίζω ότι ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε χρόνο για να απαντήσω σε κάθε μία. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν μία-μία. Αλλά όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον να τα ξανασυζητήσουμε. Είναι χαρά και τιμή για μένα να, που καλωσορίσαμε τους ε, Κροάτες συναδέλφους στην Επιτροπή σας. Ήμουν και εγώ στις επίσημες εκδηλώσεις ε, για την ε, ένταξη της Κροατίας. Ήταν θεμελιώδους σημασίας. Ήταν θαυμάσια. Δεν θα ήθελα να είμαι υπερβολικός, αλλά είχαμε όλη την εντύπωση ότι ζήσαμε μια κοσμογονική στιγμή. Υπήρξαν ε, διάφοροι συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, βουλευτές, που πήραν το λόγο. Θέλω να τους συγχαρώ όλους. Να του συγχαρώ για την επιτυχία του Άντι Μάρι στο Wimbledon. Λοιπόν, να στραφώ τώρα στα θέματα που θέσατε. Κύριε Τσαρκόφσκι. Βεβαίως. Χαιρετίζω την επικοδομητική σας τάση και τις προτάσεις σας να σας βοηθήσουμε για να βοηθηθούμε όλοι. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε. Όλοι επιδιώκουμε έναν κοινό στόχο. Όλοι θέλουμε να λύσουμε τα κοινά μας προβλήματα. για την ερώτησή σας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα γίνει η γλωσσική αναθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων θα πάρει κάποιο χρόνο Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να τελειώσουμε ε, εντός του Ιουλίου, αλλά θα σας στείλουμε το κείμενο για την επίσημη έγκριση από το Κοινοβούλιο προς το τέλος Ιουλίου, αλλά με την επιφύλαξη ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από τους ε, νομικούς λοσομαθείς και μόνο όταν δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συμφωνία του από αυτού, μόνο τότε θα μπορέσει το Συμβούλιο να το εγκρίνει επισήμως. Πολύ θίξατε το πιο σημαντικό θέμα που εκκρεμεί. που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε. συνεργαζόμενοι με την Επιτροπή σας. Το θέμα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. κάνουμε κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το δυσχερές έργο Γι' αυτό δεν έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε. Γιατί είναι δυσχερές. Έχουν γίνει διάφορες συναντήσεις για να ε, καταλήξουμε στα ε, επίμαχα ακόμη ζητήματά του, αλλά ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει. Θέλω να πω ότι η Λιθουανική Προεδρία έχει αρχίσει να εργάζεται για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι Πολύ μπορείτε να το, ορισμένοι από εσά μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Συναντηθήκαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Την πρώτη πρώτη μέρα της Προεδρίας μας. Και ήταν παρόν και ο κύριος Σεύκοβιτς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θεωρούσαμε ότι θα ήταν καλό να συναντηθούν οι επικεφαλείς των ε, τριών νομικών υπηρεσιών και ξέρω ότι θα συναντηθούν. Συναντιόνται μάλιστα σήμερα. Σήμερα είναι αυτή η συνάντηση. Για να εκπονήσουν μια πρόταση, για να ε, προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θεσμικό θέμα. Και εάν καταλήξουν σε ένα κείμενο. Θα το εξετάσουμε αύριο ήδη. Ελπίζω να καταλήξουν σε κάποιο κείμενο. Γιατί υπάρχει ένα νομικό θέμα που πρέπει να επιληθεί. Και ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουμε αρχίσει να ασχολούμεθα με αυτό. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα ποια θέματα εκκρεμούν. Είναι θεσμικής φύσης. Περιμένουμε βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση. για το πώς θα ενταχθεί το θέμα αυτό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στις εθνικές νομοθεσίες. Ελπίζω λοιπόν ότι η Κομισιό θα κάνει ε, το τμήμα της εργασίας που της αναλογεί σύντομα. Συμφωνώ και με τον κύριο Νταφ όταν λέει ότι δεν θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν εις βάρος της ποιότητας της εργασίας μας για το θέμα αυτό. Ο κύριος Χάφνερ έθεσε το πολύ σημαντικό θέμα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Λαμβάνουμε υπόψη τα σχόλιά σας, ε, κύριε Χάφνερ, για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η πρωτοβουλία αυτή. Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να επιλύσει όλες τις τεχνικές δυσχέρειες για τη συμμετοχή των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Το θέσατε πολύ. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να τα επιλύει όλα. Κατά την προετοιμασία της Λιθουανίας ε, πήγα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, συζήτησα με τους πολίτες είναι καθήκον κάθε πολιτικού. Δεν θα επιμείνω. Αλλά η Λιθουανική Προεδρία έχει σχεδιάσει πολλές πρωτοβουλίες, πολλές εκδηλώσεις για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πώς θα πιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Θέλω να επενέσω την έκθεση του κυρίου Νταφ. Και φυσικά κύριε Πρόεδρε και τη δική σας έκθεση του 2012 κύριε Καζίνη για τις προσεχείς ε, ευρωεκλογές. Καταρχάς χαιρετίζω το ότι επετέφθη συμφωνία για την ε, περίοδο των εκλογών, πότε δηλαδή θα διεξαχθούν τις ημερομηνίες των εκλογών και για την σύνθεση του Κοινοβουλίου και το μέγεθος του Κοινοβουλίου. Με συγχωρείτε τώρα, ε, σας παρακαλώ μην το πάρετε άσχημα, είναι πρώτη παρουσία ενώπιον της Επιτροπής σας. Μην το πάρετε άσχημα, μου... Επιτρέψτε μου να ξανάρθω στην Επιτροπή σας. Ε, ε, μ' αρέσει ιδιαίτερα η εργασία σας, αλλά πρέπει να αναφέρω το άρθρο 17 της Συνθήκης όπου καθορίζεται σαφώς ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για κάποιους διορισμούς, για πολύ σημαντικά αξιώματα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. για το πολύ σημαντικό θέμα της προσχώρησης της Ένωσης στην ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αλλά προς το παρόν πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου την έκθεση Μάρτενς για τις ε, εξεταστικές επιτροπές είμαστε διατεθειμένοι να βασιστούμε στην ε, επιτελεστή εργασία και θα μελετήσουμε προσεκτικά ε, τις προτάσεις που θα κάνει το Κοινοβούλιο για να επιδιώξουμε ε, την επίτευξη συμβιβασμών σε όλα τα επίμαχα θέματα. Και ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί πρόοδος για τα θέματα που, ε, όπως αναφέρει η εντολή της Κορεπέρ, δημιουργούν προβλήματα για τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, για την πρόσβαση στα έγγραφα, για τις κυρώσεις. Ξέρετε που έγκυνται οι δυσχέρειες. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε. Ο κύριος Άγνιου. Έκανε μια παρέμβαση. Προσπάθησα να μελετήσω την ε, ορολογία προετοιμαζόμενος για το καθήκον της Προεδρίας Και έμαθα λοιπόν τη λέξη ότι κάποια θέματα είναι τοξικά. Κοιτάξτε κύριε Άγνιο. Δεν με πειράζει να με απολύσουν. Εσείς θα πρέπει τι θα γίνει αν εγώ απολυθώ Γιατί στόχο μας είναι να μην χρειαστεί να απολυθώ. Είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να προωθήσουμε διάφορα θέματα. Αυτή είναι η απάντηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε μας μένει πολλής χρόνος. αλλά ε, θα επανέλθω. Έμπλεος καλής θελήσεως ενώπιον της Επιτροπής σας για να προωθήσω τα θέματα που πρέπει να επιλύσουμε από κοινό. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα σχόλιά σας, ε, τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και εύχομαι σε όλους μας κάθε επιτυχία στην προσπάθεια προώθησης των τόσο σημαντικών θεμάτων που έχουμε ενώπιόν μας τους επόμενους έξι μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την υπομονή σας που ακούσατε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε. Μα συγχωρείτε αν σας δώσαμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει αμέσως να κηρύξουμε τη λήξη αυτής της συνεδρίας γιατί ξεκινά άλλη. Άλλη για την υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να σας ευχηθώ κι εγώ ε, θερμά κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Θα έχουμε μια πολύ εντατική συνεργασία με την Επιτροπή μας και να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η πρόσημη συνεδρίαση εκτάκτος θα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Και μετά πάλι 15 και 16 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες και πάλι. Ευχαριστώ.